Wrong uh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση και το επόμενο θέμα είναι η ώρα των ψηφοφοριών. Yes. So if it is, I'd like to... Θέλετε το λόγο? Ναι, θέλω. Να θέσω ένα θέμα στα πολωνικά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα επρόκειτο να ψηφίσουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση που ε, προέκυψε μετά από τη συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία, η ε, ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Πλην όμως πριν από λίγες ώρες συνέβη κάτι ιδιαίτερο ε, ε, που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αναβληθεί η ψηφοφορία για την γνωμοδότηση αυτή skazaniu na maksymalny wyrok 7 lat więzienia. Δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια απόφαση τη στιγμή που καταδικάστηκε από δικαστήριο του Κιέβου ηγέτης της αντιπολίτευξης ε, στην ανώτατη ποινή που θα μπορούσε να δεχτεί 7 χρόνια κάθερξη. Δεν μπορούμε λοιπόν να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία δεδομένων των συνθήκων που προέκυψαν και σας καλώ να αναβάλουμε την ψηφοφορία και θα πρέπει να αποφασίσουν οι συντονιστέ και υποθέτω ότι θα ψηφίσουμε την επόμενη φορά στη συνεδρίαση της Επιτροπής μα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τι ζητάτε? Να αναβληθεί η ψηφοφορία της γνωμοδότηση για την Ουκρανία. Η γνωμοδότηση για την Επιτροπή Εξωτερικών που είναι καθήλυνα αρμόδια. Αν εμείς αναβάλουμε, κινδυνεύουμε να χάσουμε τη συνεισφορά μας αν αποφασίσει η Επιτροπή Εξωτερικών. Βεβαίως δεν μπορώ να αποφασίσω μόνος μου για αυτό το διαδικαστικό ζήτημα. Είναι θέμα της Επιτροπής, εφόσον βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Οπότε θα ανοίξει ένας πάρα πολύ σύντομος γύρος τοποθετήσεων, ένα λεπτό έκαστος συντονιστής. Η Μαρία Λιντεσαρνές πρώτη. Ήθελα απλώς να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι Συμφωνούμε απολύτως με την πρόταση του συναδέλφου Ζαλεύσκη. Θα πρέπει ε, επαόριστο να αναβληθεί η ψηφοφορία και να ζητήσουμε και από την Επιτροπή Εξωτερικών να κάνει το ίδιο. Αναβολή της ψηφοφορίας επαόριστο. Γιάννη Ξαντώ, συμφωνώ απολύτως με την αναβολή Σημειώνω ότι στη συζήτηση που κάναμε σήμερα το πρωί για μια άλλη γεωγραφική περιφέρεια, η ίδια πολιτική ομάδα μας είπε ότι θα πρέπει πρώτα να κάνουμε εμπόριο και μετά πολιτική. Εγώ υποστηρίζω αυτή την πρόταση, αλλά παρακαλώ την πολιτική ομάδα να δείχνει και κάποια συνέπεια ε, ανάλογα και με τις ε, γεωγραφικές περιοχές. Ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν ξέρουμε αν η Επιτροπή Εξωτερικών θα δεχτεί να αναβάλει και εκείνη την ψηφοφορία που είναι την άλλη εβδομάδα. Οπότε δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο να αναβάλουμε την ψηφοφορία, αλλιώ θα χαθεί η γνωμοδότησή μα. Θα έρθει κατόπιν εορτή. Οπότε, νομίζω καλά θα ήταν να ψηφίσουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στέρντι, ευχαριστώ. Υποστηρίζουμε την πρόταση και εμείς Πρόεδρε, αλλά θα πρέπει πάντα να εξετάζεται περίπτωση, να μην είναι προηγούμενο για το μέλλον. Indeed. Όντως. Οπότε, να ψηφίσουμε για το αίτημα αυτό ε, αναβολής ψηφοφορίας της νομοδότησης, είναι για την Επιτροπή Εξωτερικών. αν η ε, ΑΦΕΤ δεν μας παρακολουθήσει σε αυτή την προσπάθεια θα χάσουμε τη δυνατότητα επέμβασης στο θέμα. Α, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι θα μας ακολουθήσει και η ΑΦΕΤ. Ναι, Πρόεδρε, ο κύριος Αλεύσκη. Σήμερα συμμετείχα στη συνεδρίαση με τον Υπουργό Χουσένκο και πρέπει να σας πω ότι όλοι σχεδόν ομόφωνα εξέφρασαν έντονες επικρίσεις για τα όσα συνέφησαν νωρίτερα στην Ουκρανία. Ακριβώς την ώρα που συνεδριάζαμε παρουσία του Υπουργού, που και αυτό κάτι σημαίνει, έτσι δεν είναι. Και φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Εξωτερικών θα ε, καταλάβουν, θα σεβαστούν και θα ακολουθήσουν την απόφασή μας. Βεβαίω δεν έχω μιλήσει με όλου του συντονιστέ, με όλε τι πολιτικέ ομάδε τη Επιτροπή Εξωτερικών. Μόνο με το δικό μα συντονιστή μίλησα, που θα ζητήσει από τους συναδέλφους στην Επιτροπή Εξωτερικών να ακολουθήσουν για αυτή την απόφαση. Αλλιώς δεν θα το πρότεινα. Είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι θα μας ακολουθήσει και η Επιτροπή Εξωτερικών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την κατανόησή σας. Υπάρχει και άλλος κίνδυνος που θα ήθελα να προσθέσω. Είναι θέμα επί της ουσίας της Επιτροπής Εξωτερικών εμείς γνωδοτούμε για το εμπόριο και ενδεχομένως να μας κατηγορήσουν ότι επεμβαίνουμε σε κάτι που δεν μας αφορά, που είναι μια πολιτική εκτίμηση της κατάστασης στην Ουκρανία. Εντάξει, εσείς θα το αποφασίσετε. Να σας πω κι εγώ την προσωπική μου άποψη, δεν θέλετε. Ο Καντέρα Ρίφ. Να τελειώνει η συζήτηση. Ναι, ναι, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετική ε, αντίληψη. βεβαίως και το εμπόριο πολιτική υπόθεση είναι. Ξέρετε ότι εγώ δεν θεωρώ ότι το εμπόριο είναι αμυγός τεχνικό θέμα. Ε, σημειώνω αυτό που είπε ο Γιάννη Ζαντό, ότι δεν μπορούμε να επιλέγουμε. Παρόλο που είναι πονηρός ο Ρόμπερτ Στέρντι, δεν θα πρέπει να κάνουμε διάκριση αναπεριοχή. Ε, καταρχήν ε, είμαι υπέρ λοιπόν της ε, αναβολής και υπέρ της πρότασης του συναδέλφου Ζαλεύσκη. Εντάξει, ψηφίζουμε, λέει ο Πρόεδρος, ψήφι υπέρ της αναβολής αυτό που ζήτησε ο Αντιπρόεδρος Πάβελ Ζαλεύσκη αναβάλλεται η ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση για τη συμφωνία με την Ουκρανία. Σαφής η πλειοψηφία κατά αποχές σαφής πλειοψηφία υπέρ αναβάλλεται η ψήφιση της γνωμοδότησης για την Ουκρανία. Τα υπόλοιπα που πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Σημείο 11. Ο εισηγητής, για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου ζητεί να κάνει πρόταση η Επιτροπή μας στο Κοινοβούλιο να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως προς το, νόμιμο, το νομότυπο της συμφωνίας αυτή. Θυμίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 6 του κανονισμού uh, που εφαρμόζει πλέον ε, το γράμμα της συνθήκης. Πριν ψηφίσουμε ε, για τη σύμφωνη γνώμη σε μια διεθνή συμφωνία, κάποιος, ε, μια πολιτική ομάδα ή ένα δέκατο των μελών μπορεί να ζητήσει το Κοινοβούλιο να προσφύγει στο ΔΕΚ προδικαστικά, μάλλον να κάνει μια αίτηση για ένα ερώτημα για τη συμφωνία αυτή. Λοιπόν, το Κοινοβούλιο συμμετέχει με δύο τρόπους στην ψηφοφορία ε, για τη Διεθνή Συμφωνία και για την προσφυγή στο ΔΕΚ. Είτε με ένα δέκατο λοιπόν των μελών, είτε ε, μια πολιτική ομάδα, είτε μια επιτροπή. Εμείς επιτροπή είμαστε και ένα μέλος της επιτροπής ζητεί ε, να ζητήσει η Επιτροπή μας από το Κοινοβούλιο να προσφύγει στο ΔΕΚ. Uh, ε, προσφύγουμε στο δικαστήριο για αυτό το θέμα. Το καταλάβαμε λοιπόν, θα πρέπει να ψηφίσουμε. Είστε υπέρ του αιτήματο του κυρίου Ζωζέ ή όχι. Μου ζήτησε ο εισηγητή να το επιτρέψω να εξηγήσει τους λόγους που τον εκκίνησαν να κάνει αυτή την πρόταση. Παρακαλώ, τρία λεπτά κύριε Μποβέ για να εξηγήσετε τη θέση σας. Παρακαλώ. Merci, euh, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που εγγράψατε στην ημερήσια διάταξη αυτό το αίτημά μου και που υπενθυμίσατε το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Γιατί πρότεινα να γίνει αυτό σε επίπεδο επιτροπής. Γιατί είναι ένα θέμα δικαίου και όχι πολιτικό ζήτημα που θα έθεταν ενδεχομένως 75 βουλευτές ή μια πολιτική ομάδα. Δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι θέμα νομικό. Έτσι. Το πρώτο σημαντικό να θυμίσουμε, το ΔΕΚ θεωρεί ότι οι αρμοδιότητες της Ένωσης θα πρέπει να ασκούνται ε, ε, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και αυτοί οι κανόνες είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωμης Τάξης. Αυτό είναι σημαντικό. Έχω κάποιες επιφυλάξεις όμως ε, στη συμφωνία αυτή που έχουν να κάνουν με το ειδικό ιδιαίτερο καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας σε σχέση με την Ισπανία αφενός που νομικά είναι υπεύθυνη και το Μαρόκο αφετέρου που είναι de facto υπεύθυνο και όχι de jure. Αν δούμε τα κείμενα λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών, σήμερα ξέρουμε ότι το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας δεν έχει ξεκαθαριστεί και σε σχέση με το μέλλον ε, ε τη επικράτησης αυτή ε, η προσπάθεια. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πολιτικό να δούμε πού γέρνει η πλάστηγκα αν είμαστε δηλαδή με το Μαρόκο ή ε, με κάποια άλλη πολιτική ε, δύναμη που θα πρέπει να χειρίζεται και να διαχειρίζεται την επικράτεια αυτή. Ε, το μόνο που μας απασχολεί είναι να μπορεί να ενταχθεί σε μια συμφωνία διεθνή. Το σχέδιο όμως που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σήμερα εμεί καλούμε θα να υπάρχει μια μεγάλη αδυναμία δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να επιτρέπει να λέμε εάν ναι ή όχι η Δυτική Σαχάρα είναι εντός της περιμέτρου ε, της συμφωνίας. Αν είναι εκτός της συμφωνίας καλός, αν είναι εντός όμως όπως έχει ακουστεί επανειλημμένα, είδαμε και άλλες χώρες και θυμίζω τις Ηνωμένε Πολιτείε διαστόματος Ρόμπερ Ζέλικ που σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν κάνει διαφοροποίηση στη Συμφωνία εταιρική σχέση. Από τη μία είναι το Μαρόκο λοιπόν και από την άλλη είναι αυτά τα εδάφη, τα μη αυτό όνομα της Δυτικής Σαχάρας. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το θέμα να το ε, ξεκαθαρίσει ένα δικαστήριο ε, εάν υπάρχει συμβατότητα όχι και σας ζητώ χωρίς καμία πολιτική φόρτιση χωρίς ε, να σκέφτομαι τίποτα διαφορετικό με τρόπο πάρα πολύ νυφάλιο και ήρεμο να το λύσει αυτό το θέμα το δικαστήριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τι θα ψηφίσουμε, να είμαστε σαφείς. Εάν ψηφίσουμε ναι τώρα σε αυτό που θα σας ζητήσω, ζητούμε από το Κοινοβούλιο να προσφύγει στο δικαστήριο. Εάν ψηφίσουμε όχι, δεν θα γίνει. Καντέρα Ρίφ. Καντέρα το Καντέρα Ρίφ. Πρόεδρε, θέλω να θέσει υπόψη των συναδέλφων την απόφαση, σοφή θεωρώ, των συντονιστών σήμερα το πρωί για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Ε, ζητείτε διευκρίνηση για πολλά θέματα, όχι μόνο για τη Δυτική Σαχάρα και η αναβολή αυτή η καθυστέρηση μάλιστα θα έλεγα και η προθεσμία που θα μας επιτρέπει να μπούμε στην ουσία με ακρόαση ενδεχομένως όπως αποφάσισαν σήμερα το πρωί οι συντονιστές και νέα ακρόαση για να προσπαθήσουμε να έχουμε περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν με κάνουν να πιστεύω τα εξή. Πρέπει να ψηφίσουμε για την προσφυγή στο ΔΕΚ σήμερα. Είναι απαραίτητη η ψηφοφορία. Ε, Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι την ακρόαση να έχουμε περισσότερη ενημέρωση ε, και όχι απλώς με μια απλή ψηφοφορία ναι ή όχι για προσφυγή στο δικαστήριο. Είχαμε αποφασίσει, αποφασίσαμε στους συντονιστές να το αναβάλουμε για ένα μήνα το θέμα αυτό αντί να έχουμε το πρώτο, το πρώτο προσχέδιο που θα εξετάσουμε, την πρόταση ψηφίσματος δηλαδή το Νοέμβριο και την ψηφοφορία το Δεκέμβριο, αποφασίσαμε να αναστείλουμε για ένα μήνα, το οποίο σημαίνει θα εξετάσουμε το σχέδιο πρότασης το Δεκέμβριο και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει τον Ιανουάριο. Αυτό αποφασίσαμε αυτή τη μετατόπιση δηλαδή, τη χρονική και έτσι προσαρμόσαμε και το χρονοδιάγραμμά μας. Άρα θα αποφασίσετε εσείς κατά πόσο υπάρχει αντίκτυπος του χρονοδιαγράμματος σε σχέση με την ενδεχόμενη προσφυγή στο ΔΕΚ. Αυτή είναι μια πρόταση αναστολής της ψηφοφορίας. Εγώ θα... Εσείς θα το αποφασίσετε, δεν μπορώ να το αποφασίσω εγώ. Κασπάρη, αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δική μας πρόταση του ΕΛΚ να προσφύγουμε τώρα στο δικαστήριο. Ο εισηγητής το ζήτησε. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Και μεταξύ άλλων, γιατί ο εισηγητής καθυστερεί αυτό το θέμα εδώ και μήνες, δεν τηρεί κανένα χρονοδιάγραμμα και αν ήθελε να λυθεί κάτι, να ρωτούσαμε τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλα αυτά τα πράγματα δεν συνέβησαν, δηλαδή τον εισηγητή δεν τον ενδιαφέρει να βρεθεί κάποια λύση κατά την άποψή μου παρά μόνο να χρονοτριβεί και να η εργή και παρακαλώ να ψηφίσουμε και άμα θέλει να απευθυνθεί στην νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου να το κάνει άλλη στιγμή. Να ψηφίσουμε την έκθεση λέω. Ακούσαμε μία γνώμη κατά, έχουμε υπέρ κανέναν, όχι. Υποτεθέτω ότι δεν υπάρχει υποστήριξη για την αναβολή της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Please, uh, what about your cards? And the vote is... Πέρασε. Της ψηφοφορίας 26 ψήφισαν από τους 29. The vote is closed. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Με 19 ψήφους κατά, 5 υπέρ και 2 εποχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ας προχωρήσουμε στο σχέδιο έκθεσης. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία, λέει ο Πρόεδρος. report on trade and investment φραγμή στο εμπόριο και επενδύσεις του εισηγητή, του κυρίου Στέρτη. Θέλει κάτι να μας πει ο εισηγητής. Ευχαριστώ καταρχήν. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες και το προσωπικό τους για να φτάσουμε σε συμβιβασμού, σε προτάσεις συμβιβασμού. Υπάρχουν πολλές ε, τροπολογίες, από 64 φτάσαμε σε 13 προτάσεις συμβιβασμού με μία ή δύο εξαιρέσεις. Δεν είμαστε η αρμόδια αρχή και δεν μπορούμε να αποφανθούμε σε συγκεκριμένες περίπτωσεις, ιδιαίτερα ως προς τις, τους φραγμούς στο εμπόριο. Γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν διαφορές και αυτό αντικατοπτρίζει και τις συζητήσεις που είχαμε με την Επιτροπή στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Οι τροπολογίες μιλούν για αριθμιστικής μορφής διάλογο με τους στρατηγικούς εταίρους και συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούνται αυτοί οι, εμπορικοί, οι μη εμπορικοί φραγμοί. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προβούμε σε μία διάκριση μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών και αναδυόμενων οικονομιών, δηλαδή χωρών BRIC, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρώτες ύλες ή δασμούς κατά τις εξαγωγές. Στην περίπτωση της Ιαπωνίας και ως προς τα διεθνή πρότυπα υπάρχει μια ξεχωριστή πρόταση, αλλά το δικό μας κείμενο αποτιμά σωστά το θέμα. Εάν εγκριθεί η έκθεση και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν από, όλο το πολιτικό φάσμα και πιστεύω ότι θα πρέπει να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα ε, συντάξει τη δική της έκθεση το Μάρτιο. Ωραία. Ας αρχίσουμε τις πληροφορίες. Πέντε σελίδες έχουμε. 64 τροπολογίες. Ας αρχίσουμε με το συμβασμό υπαριθμών 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ... Α, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Καταπίπτει το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Υπάρχουν αμφιβολίες, θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, 21 τμήμα 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. And vote is closed. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία... Μάλλον τροπολογία συμβασμού 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σοβαρολογείτε, θέλετε να ελέγξουμε, ωραία. Ελέγχουμε την 27. 28. 27. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές, δεν είμαι και τόσο σίγουρος, ας ελέγξουμε. Την 28 αρχίζει η ψηφοφορία. Εντάξει, τώρα λειτουργούν τα μηχανήματα, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας, ισοψηφία απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 ελέγχουμε αφού το θέλετε. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 30. What post? Απορρίφθηκε. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Ωραία, ας ελέγξουμε και την 31. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβασμού 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβασμού 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ω, να ελέγξουμε, θέλετε να ελέγξουμε, εντάξει, 42 ελέγχουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. 42, 42, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. The Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία συμβιβασμού 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία συμβιβασμού 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία συμβιβασμού 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 54. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 και 56 είναι παρεμφερείς υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία συμβιβασμού 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβασμού 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Μόνο το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχοντας υπόψη η τροπολογία συμβασμού 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία συμβασμού 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβασμού 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. 7 και 8 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία συμβασμού 4. Ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Θέλετε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας συμβασμού 4. Δεύτερο τμήμα, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 13. 13. Τροπολογία 13. Αμε συγχωρείτε. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα αιτιολογικές σκέψεις 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι τροπολογίες της ΣΥΜΚΟ 7. Υπαριθμών 7 της ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 10 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Ήμκο 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. And vote is closed. Πέρας. Και εγκρίθηκε με 23 ψήφους υπέρ, 4 κατά. Να συγχαρούμε τον εισηγητή μας για την ε, επιτυχή αυτή έκβαση. Θέμα 13. Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότησης της Κριστιάνα Μουσκαρντίνη Θα πρέπει να σας πω ότι η κυρία Μουσκαρντίνη έπεσε, έσπασε το χέρι της, βρίσκεται στο νοσοκομείο και ζήτησε συγγνώμη γιατί δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Εξ ονόματος όλων λοιπόν, τις εύχομαι... Μπορούμε να στείλουμε και λουλούδια, λέει κάποιος. Τις εύχομαι καλή ανάρρωση. Θα το ρυθμίσω, λέει ο πρόεδρος. Δεκατέσσερις υπέρ, 15 ε, υπέρ μάλλον, με μία ψήφο παραπάνω, θα θέλαμε να σε ευχηθούμε καλή ανάρρωση. Λοιπόν, έκθεση Μουσκαρδίνη. Σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, τροπολογία συμβιβασμού 1. Υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίθηκε. Τροπολογία συμβιβασμού 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 11. 11 και 2. Αν θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε την 10. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Με συγχωρείτε γι' αυτό. 11 και 12 μαζί, γιατί είναι παρόμοιες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Α, δεν ψηφίζουμε. Με συγχωρείτε. Πρόκειται για ένα συντακτικό γλωσσικό θέμα. 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά Ας επαναλάβω, 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίθηκε με 24 ψήφους υπέρ 4 και 0. Λοιπόν, προχωράμε στο 15, γιατί το 14 το έχουμε αναβάλει για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Άρα ψηφίζουμε το 15 για τη Γεωργία. Συμφωνία Σύνδεσης με τη Γεωργία της κυρίας Αντρικένε. Και αρχίζουμε με την τροπολογία συμβάσμου 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού, όχι με συγχωρείτε, 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε την 9. 9. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία συμβιβασμού, λέει ο πρόεδρος και σταματάει και διακόπτει. Μα δεν, ε, ε, δεν φέρατε αντιρρήσεις εν γέρος. Τέσσερα υπέρ. Τροπολογία συμβιβασμού τέσσερα υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβασμού 5. Υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε 22 υπέρ 3 κατά και δύο αποχές. Να συγχαρούμε και πάλι την εισηγήτρια, την κυρία Αντρικένε. Φτάσαμε στο τέλος της ώρας ψηφοφοριών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Γρήγορα τα καταφέραμε. So we And please, don't get excited. Σας παρακαλώ, ησυχάστε λίγο. We are doing our job. Δεν θέλω υπερδιέγερση. Θέλετε να διακόψουμε για λίγο, για πολύ λίγο. Όσοι είναι να αποχωρήσετε, κάντε το σύντομα. And quietly not have in this room. Χωρίς συζητήσεις και πηγαδάκια εντός. Εκτός, ευχαρίστως. Κάντε ό,τι θέλετε. May I have your attention, please? Thank you. We have now a hearing um, on... Λοιπόν, αρχίζει η ακρόασή μας και το θέμα είναι η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Ε, ανισομέρεια στο εμπόριο. Η κυρία Σαρνέζ είναι η συγγήτριά μας. Δε Σαρνέζ, δε Σαρνέζ. Πού είναι το πρόγραμμα, αναρωτιέται ο πρόεδρος, το αναζητάει και περιμένουμε. I have here the program. So let's start. Το κάνεις να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 Maybe continue. Okay, Ladies and gentlemen, Κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε τη δουλειά λοιπόν. Έχουμε μια ακρόαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα και η ερώτηση είναι ασύμετρο εμπόριο, μη ισορροπημένο εμπόριο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα. Η Κίνα έχει επαναδειθεί ως η μοναδική ενιαία οικονομία στον κόσμο. Οι εμπορικέ σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια δραματικά. Η ε, Κίνα είναι ο δεύτερο ε, εμπορικό εταίρο μετά τη ΗΠΑ και ε, ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών. Επίσης, η ε, ΕΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της, της Κίνας και αυτό έχει ε, αυξήσει ε, τα, τις από την Κίνα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να ανοίξει εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. Αυτή τη στιγμή το εμπόριο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα έχει μεγάλο έλλειμμα για, έλλειμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν ανησυχίες ε, με την, σχετικά με τη συμμόρφωση της ε, Κίνας με τους κανόνες του ΟΠΟΕ σχετικά με την προστασία των ε, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης υπάρχουν θέματα περιβάλλοντος τα οποία έχουν γερθεί και επιπρόσθετα η Κίνα ε, χρησιμοποιεί, λέγεται ότι χρησιμοποιεί το, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για να αυξήσει τις εξαγωγές. Εδώ θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση εις βάθος για το θέμα προτού συνταχθεί η έκθεση και γι' αυτό το λόγο έχουμε καλέσει ε, ορισμένους εξωτερικούς εμπειρογνώμονε για να δώσουν τη δική τους παρουσίαση και να συμμετέχουν στην Σύνοδο Ρωτοκρίσεων μαζί με τα μέλη της Επιτροπής. Και χαίρομαι πολύ να παρουσιάσω εδώ ενώπιόν σας ε, τους διακεκριμένους εμπειρογνώμονές μας. Δυστυχώς ο κύριος Άντριου Γου, ο διευθυντής ε, του ομίλου Louis Vuitton Met Hennessy στην Κίνα ε, επέστρεψε επιγόντως στη Σανχάη σήμερα από το ταξίδι στην Ευρώπη και ε, έχει ε, ζητήσει συγγνώμη για την απουσία του εδώ στην Επιτροπή. Οι εμπειρογνώμονες που είναι παρόντες είναι η κυρία Λέιλα Σουκρούν Μπορεί να μην προφέρω σωστά τα ονόματά σας, λέει ο Πρόεδρεύων. Ε, υπεύθυνη για ε, την, έκθεση που έχει ανατεθεί από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Γιώνας Παρέλο Πλέσνερ. ο οποίος είναι ανώτερος υπεύθυνος πολιτικής στο ECFR Λονδίνου, ο κύριος Αντουάν Μπρουνέ, πρόεδρος της AB Marché από το Παρίσι, ο κύριος Τζόναθαν ε, Χόλσλαγκ, επικεφαλής της έρευνας στο ε, Βρετανικό Ινστιτούτο Σύγχρονων Κιναζικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο ε, VUB στο Βρυξέλλες, ο κύριος Βιωρέλ Πιστιτσάια Μπουντούρα Με συγχωρείτε για την κακή προφορά του ονόματός σας, λέει ο Πρόεδρος. Ε, διευθύνων Σύμβουλος EEAS Ασία στην έδρα τους εδώ στις Βρυξέλλες. Και η κυρία Χέλενα Κένι, ε, επικεφαλής της μονάδας ε, στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για τις σχέσεις με την Κίνα. Θα ήθελα να δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στην Μαριέλ Ντεσαρνές, που είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπατε. Πολύ σωστά, εν είδη εισήγησης. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τους παρόντες γιατί όλοι ο καθένας στον τομέα του είναι ε, ε πανεπιστημιακός, διανοούμενος, εμπειρογνώμονας, ε, γνωρίζει τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις Ευρώπης-Κίνας και θα ήθελα να τους ακούσουμε πριν, επειδή έχουμε καθυστερήσει αρκετά, γιατί εκείνους θα πρέπει να ακούσουμε σήμερα και μετά θα προβούμε σε ένα διάλογο, δηλαδή μεταξύ εμπειρογνωμόνων και μελών και μετά θα φτάσουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αυτό προτείνω, Πρόεδρε. Ναι, βεβαίως, ευπρόσδεκτα αυτά τα σχόλια. Ας ακούσουμε, ας αρχίσουμε να ακούμε τους ε, εμπειρογνώμονες και θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Λέιλα Σουκρούν να μας κάνει την παρουσίασή της. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους εμπειρογνώμονες να μην υπερβούν τα δέκα λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέγομαι Λέιλα Σουκρούν, είμαι καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μάστριξ στην ε, Σχολή Νομικής και είναι μεγάλη τιμή μου και χαρά μου που σας παρουσιάζω ε, αυτή την μελέτη Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα Ανισομέρεια στο Εμπόριο που έγινε από μια ομάδα μελετητών στο Πανεπιστήμιο του Μάστρικ και στο London School of ε, Economics και την οποία συντόνισα εγώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να παρουσιάσω τη δομή της μελέτης μας. Όπως βλέπετε έχουμε πέντε κεφάλαια μιας περιεκτικής μελέτης για τις ε, εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας με εστίαση κυρίως στους εμπορικούς φραγμούς και την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τον ΠΟΕ της Κίνας έχουμε το θαύμα της Κίνας ή ε, απειλή της Κίνας. Η Κίνα είναι στο επίκεντρο κάθε οικονομικής συζήτησης σήμερα και περισσότερο από ποτέ ε, θεωρείται ως ένα στρατηγικά σημαντικός εταίρος. Μια πρόσφατη μελέτη από το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο στην Κίνα δείχνει ότι 78% των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν έχουν ε, κέρδη στην Κίνα και 71% αναφέρουν καθαρή αύξηση σε αυτά τα κέρδη. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές εταιρείε έχουν εκφράσει κάποιες ανησυχίες για το αυτό που αποκαλούν ένα ανισομερέ επίπεδο συνεργασία με την Κίνα. Οι ευρωπαϊκές εταιρείε είναι πολύ ευαίσθητε στην περιπλοκότητα και την μη διαφάνεια του ρυθμιστικού πλαισίου στην Κίνα. Δέκα χρόνια μετά από τη δραματική ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ, αυτό γύρει μια σειρά πολύ σημαντικά ζητήματα σχετικά με τη ε, δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά ε, από τις ευρωπαϊκές εταιρείες και επίσης για την ελκυστικότητα της κινέζικης αγοράς που θεωρείται στρατηγικώς δύσκολο να διεισδύσει κανείς. Θα ήθελα να αναπτύξω αυτό το θέμα. Από το 1989 μέχρι σήμερα οι ε, εμπορικέ σχέσει Κίνα-Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σημαντικά ε, βελτιωθεί. Αλλά η κατάσταση είναι κάπως θεταμένη. Η οικονομική κράση φυσικά και η κρίση του δημοσίου χρέους επίσης έχει οδηγήσει στην επιδίνωση ε, αυτών των εντάσεων. Αφενός έχουμε μια ε, Κίνα η οποία είναι λιγότερο πρόθυμη να δεχτεί συμβιβασμούς σε διεθνείς ε, εμπορικές διαπραγματεύσεις. Το βλέπουμε αυτό σε επίπεδο του ΠΟΕ. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε κλήσεις για περισσότερο προστατευτισμό που έχουν εγερθεί σε ευρωπαϊκέ χώρες, σε ευρωπαϊκού κύκλου, γενικά. Αυτέ οι εντάσει έχουν οδηγήσει στο ε, να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια ισχυρή θέση απέναντι στην Κίνα ε, και παρόλο που οι πολιτικές ε, σχέσεις παραμένουν καλές θα λέγαμε. Είναι ενδιαφέρον για μας γιατί οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας μπαίνουν σε μια νέα φάση. Πριν από 30 χρόνια, και είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας, πριν από 30 χρόνια η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν δεν είχαν καθόλου εμπορικές σχέσεις. Βεβαίως οι εμπορικές σχέσεις έχουν ε, αυξηθεί δραματικά. Ιδιαίτερα μετά το 2002-2003, κατά τελευταία δεκαετία το εμπόριο σε αγαθά ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα έχει αυξηθεί κατά 400% από το 2007 η Κίνα έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών. Αλλά όλοι το γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα διαρθρωτικό έλλειμμα από το 1997 με τα αγαθά της Κίνας. Αυτό το έλλειμμα είναι 26 φορές μεγαλύτερο από το εμπορικό πλεόνασμα στις υπηρεσίες. Κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει πλεόνασμα εμπορικό με την Κίνα. Αλλά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχει κανείς κατά νου, αλλά λέω, αυτό το εμπορικό έλλειμμα οφείλεται στην επανεξαγωγή την Ευρωπαϊκή Ένωση αγαθών που παράγονται από ευρωπαϊκέ εταιρείε και τι δικατρικέ του στην Κίνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τι επενδύσει, η κατάσταση είναι κάπω διαφορετική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το προβάδισμα απέναντι στην Κίνα. Θα ήθελα να ε, απευθυνθώ στο θέμα ε, της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Κίνα απέναντι στον ΠΟΕ. Εδώ η περιπλοκότητα και ε, εξαιρετικός χαρακτήρας του πρωτοκόλου πρόσβασης της Κίνας στον ΠΟΕ ε, χρήζει προσοχής. Το πρωτόκολλο ε, ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ είναι μοναδικό γιατί ενσωματώνει ε, κάποιες δεσμεύσεις ΠΟΕ συν σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις ΠΟΕ πλην η Κίνα, σε αντίθεση με όλα τα άλλα μέλη, έχει αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις παραδοσιακές, αλλά και κάποιες μη παραδοσιακές υποχρεώσεις του ΠΟΕ. Άρα, οι δυσαρέσκειες ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή του πρωτοκόλου ένταξης της Κίνας θα πρέπει να θεωρηθεί σε ε, συνδυασμό με τον μοναδικό χαρακτήρα αυτού του πρωτοκόλου. Επιπρόσθετα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε, ε, αυτές, ε, κάποιες από αυτές τις υποχρεώσεις μέσα στο πρωτόκολλο για να μην μιλήσουμε και για την απουσία οποιασδήποτε δικαιολόγησης για την επιβολή κανόνων που παρεκκλίνουν από τους γενικούς κανόνες μη διάκρισης είναι αμφισβητήσιμα. Μπορεί να δει κανείς μια πιο δυνατή Κίνα που μπορεί να υπεραμεινθεί κατά ε, πολλών δεσμεύσεων που θεωρεί άδικες και να παίζει ένα πιο προενεργητικό ρόλο και να κάνει μια πιο προενεργητική χρήση του συστήματος επίλυσης διαφορών ε, στον ΠΟΕ. Η μελέτη μας έχει ε, δώσει πολλές πληροφορίες για τους εμπορικούς φραγμούς, ιδιαίτερα φραγμούς στο ε, στο σύστημα αλλά και το, το θέμα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ε, βιομηχανική πολιτική της Κίνας και επίσης στον τομέα της γεωργίας. Υπάρχει ένα τμήμα για τους εμπορικούς φραγμούς που εστιάζεται κυρίως στο θέμα της μεταβίβασης τεχνολογίας, ε, των, της διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλων θεμάτων. Για την εκτέλεση της μελέτης χρησιμοποίησαμε φυσικά τις πρόσφατες αναθεώρησεις σε επίπεδο ΠΟΕ ε, μέσα στον, ε, και επίσης τον μηχανισμό αναθεώρησης της ε, πολιτικής, εμπορικής πολιτικής και έχουμε δει επίσης και άλλες μελέτες που έχει διενεργήσει η Αμερικανική κυβέρνηση. Θα πρέπει να πούμε ότι παρόλο που κάποιες πηγές υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει συντονισμός και δεν είναι πάντα τόσο χρήσιμες όσο θα ανέμενε κανείς. Τώρα για να συνοψίσω γιατί βλέπω ότι δεν έχω πολύ χρόνο και θα ήθελα να κάνουμε και μια οικοδομητική συζήτηση. Θα δώσω κάποια ε, καταληκτικά λόγια τώρα και θα έλεγα ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, είναι καλά εξοπλισμένες για να υπερπηδήσουν και να ε, ξεπεράσουν αυτή την πρόκληση της Κίνας. Αλλά θα πρέπει να υποστηρίζονται από μια ευρωπαϊκή πολιτική που να κατευθύνεται ακριβώς στα προβλήματα της Κίνας. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια σταθερή θέση για να ξεπεράσει αυτό τον κατακαιρματισμό που παρατηρείται σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για όλες τις ερωτήσεις. I uh, Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ακούσουμε τώρα στον ε, κύριο Γιώνας Παρέγιο Πλέσνερ, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις εξωτερικές σχέσεις. Που είσαστε εδώ μπροστά σας. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή με τιμά ιδιαίτερα, όπως είπατε και εσείς, η Κίνα έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους πολίτες και για τις χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η σύγκληση αυτής της ακρόασης. Εγώ προέρχομαι από το Think Tank που αφορά τις ε, εξωτερικές σχέσεις. Είναι το μόνο πανευρωπαϊκό Think Tank το οποίο ασχολείται με θέματα ε, εξωτερικών υποθέσεων. Μεταξύ αυτών μας απασχολεί και η Κίνα. Εξετάζουμε και τις σχέσεις μας με την Κίνα. Θα προσπαθήσω, μια και έχω μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μου, να ασχοληθώ με ορισμένες συστάσεις για το πώς η Ευρώπη θα μπορούσε να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Κίνα ένα συνάδελφος, ο Φρανσουά Γκουτμάν, συνέταξε αυτή την ε, έκθεση που σας δείχνω σε σχέση με τη νέα οικονομική παρουσία της Κίνας στην Ευρώπη και έτσι έχετε μία σχετική εικόνα. Στη συνέχεια θα μιλήσω για τις συστάσεις αυτές για να τις εντάξουμε στη συζήτηση. Η ευρωπαϊκή κρίση αποτελεί ευκαιρία για την Κίνα γιατί λίγο καιρό πριν οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Κίνας αφορούσαν φθηνές εξαγωγές ή εισαγωγές της Κίνας, στη, της Κίνας στην Ευρώπη. Τώρα όμως αλλάζουν οι συσχετισμοί δυνάμεων. Πέρσι το μεγάλο κουαρτέτο, ο πρόεδρος Γου και ο πρωθυπουργός, ο Σιαν Λί, και ένας άλλος οικονομικός ε, ιδίμων έκαναν ένα γύρο από τις ευρωπαϊκές, ε, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στη Λισαβόνα, στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, για να αλλάξει η οπτική γωνία, μάλλον η αντιμετώπιση της Ευρώπης ως προς την Κίνα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρώην κομμουνιστικό σύστημα ήταν ιδιαίτερα δύσπιστο ως προς την Κίνα. Και ο Βίκτορ Όρμπαν, ο ε, Πρωθυπουργός, υποδέχτηκε τον Δαλάι Λάμα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όταν ο Δαλάι Λάμα λοιπόν έκανε αυτή την επίσκεψη και ο Όρμπαν επανήλθε στην εξουσία, Τότε κανένας δεν τον υποδέχτηκε και φέτος ο Πρωθυπουργό Βουέγγ μας μιλούσε για τον ιστορικό αυτό, τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Ουγγαρίας και Κίνας. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν συσχετισμοί δυνάμεων και αντιλήψεων που αλλάζουν άρδιν και πολύ γρήγορα. Επίσης η Ευρώπη θα προωθήσει την ε, αρρωγή προς την Κίνα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η Κινέζικη Τράπεζα Ανάπτυξης ε, διευρύνει τις σχέσεις της προς την Ευρώπη. Και αυτό αποτελεί μια άλλη σημαντική αλλαγή. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς μπορεί η Ευρώπη να ενταχθεί στη στρατηγική της Κίνας και τι αποζητά η Κίνα. Αν λοιπόν κοιτάξουμε το επόμενο πενταετές ε, πρόγραμμα, βλέπουμε ότι η Ευρώπη εντάσσεται πολύ καλά διότι η Κίνα θέλει να κινηθεί προς την πράσινη ανάπτυξη, προς μια αναδυόμενη οικονομία, αναπτυσσόμενη οικονομία και σε επενδύσεις προς την Ευρώπη. Αυτό το βλέπουμε και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Βλέπετε ότι η που έχει περάσει στην κινέζικη Μπετζίλη και βλέπουμε ότι θα υπάρξει και κάποια συνέχεια. Και το ίδιο θα ισχύσει και για τη ΣΑΜΠ. Επίσης υπάρχουν μονάδες κατασκευής αυτοκινήτων πλέον στη Βουλγαρία. Όταν μιλάμε για επενδυτικά σχήματα θα πρέπει να, να μην ξεχνάμε ότι ότι αρχικά οι επενδύσεις ήταν πολύ χαμηλές, αλλά τώρα έχουν επιταχυνθεί. Και το ίδιο αφορά ε, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Επίσης, ως προς επενδύσεις της ΕΠΑ είδαμε ότι στο 2020 θα έχουν ανέλθει σε ένα τρεις και μέσα στα πλαίσια του πενταετούς προγράμματος θα γίνει λόγος για εξαγορές προϊόντων τεχνολογίας εχμής και μέσα στη στοχοθέτηση αυτή εντάσσεται και η Ευρώπη. Και αυτό αφορά την γενικευμένη κρίση που ισχύει όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ. Επίσης, η Κίνα θέλει να μπορέσει να καταθέσει κεφάλαιο στις τράπεζες του εξωτερικού και βλέπετε λοιπόν ότι και η μεγάλη μας κρίση στον τραπεζικό τομέα θα μπορούσε να προσελκύσει τους Κινέζους. Αυτό αφορά και τα σχέδια ιδιωτικοποίησης που γνωρίζουν η Πορτογαλία και η Ελλάδα ιδιαίτερα που ενδιαφέρουν τους Κινέζους. Δεν θα πρέπει να κατηγορήσουμε την Κίνα γιατί θέλει να δράξει αυτή την ευκαιρία. Ο υφυπουργό εξωτερικών, ο Φου Γιέγκ, είχε ε, ε, πει ότι είτε αγοράσουμε είτε δεν εξαγοράσουμε, δηλαδή είτε κάνουμε εξαγορές είτε όχι, οπωσδήποτε θα μας δακτυλοδεικτούν, έτσι κι αλλιώς, θα μας κατηγορούν. Άρα οι Κινέζοι θέλουν να δαπανίσουν και να επενδύσουν τα χρήματά τους και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς εμείς συλλογικά ως Ευρωπαίοι μπορούμε να ε, έχουμε ευεργετήματα από αυτή την κατάσταση προς την κρίση της Ευρώπης, τη χρηματοπιστωτική ε, κρίση και την εξαγορά του χρέους έχει αποστείλει μηνύματα στην Ουγγαρία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Έχει αποστείλει σήμα προς αυτές τις χώρες η Κίνα ότι θέλει να εξαγοράσει ένα μέρος του χρέους. Γίνεται λόγος λοιπόν για εξαγορά ενός μέρους του χρέους αυτών των χωρών, αλλά αυτή η εξαγορά θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και τη στιγμή που η ΕΚΤ και το EFSF προβάλλουν τα δικά του σχέδια, η Κίνα δεν μπορεί να ενταχθεί πάντα σε αυτά. Η Κίνα με τα ε, μεγάλα αποθέματα μπορεί να αλλάξει και να αγοράσει ομόλογα τριπλού α και αυτό αφορά αγορές κυρίως από την, ε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Γερμανίας. Επίσης ε, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο διότι ως προς τα δημόσια ομόλογα και την εξαγορά τους δεν είναι ξεκάθαρη κατάσταση και οι πολιτικοί δεν ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Υπάρχουν θέματα λοιπόν των, εμο, των ευρωμολόγων και των ομολόγων ε, γενικότερα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη ΣΥΠΑ έχουμε τα στοιχεία GHE τα οποία είναι εντελώς διαφανή και μπορεί να τα λάβει κανείς από οπουδήποτε θέλει. Το ίδιο δεν ισχύει για την Ευρώπη και το δημόσιο χρέος της, ε, ιδιαίτερα ως προς τις αγορές της Σανγκάης και του Χονγκ Κονγκ. Άρα τα πράγματα δεν είναι πάντα ξεκάθαρα. Ως προς επενδύσεις, οι κινέζικες επενδύσεις είναι πολύ καλές και προς την Ευρώπη αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κάνουν ανοίγματα προς την Κίνα. Ενώ λοιπόν η Ευρώπη παραμένει ανοιχτή στις επενδύσεις, το Πεκίνο προβάλλει στάση προστατευτισμού έναντι των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεών της. Δηλαδή δεν είναι πάντα αμφίδρομη αυτή η πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει ένα σύμφωνο εμπορικών σχέσεων, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλείς επενδύσεις και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Κίνα και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Έτσι ώστε ως προς τα προϊόντα τεχνολογίας εχμής δεν θα πρέπει να πρόκειται για μια καθαρά εγχώρια κινέζικη αγορά, αλλά να έχουν πρόσβαση και οι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν θέμα ασφάλειας και διαφάνειας διότι πολλές φορές οι επενδύσεις, τις επενδύσεις διαχειρίζονται κρατικοί φορείς. Και εδώ υπάρχουν πολιτικά καθαρά συμφέροντα. Εδώ χρειάζεται απόλυτη διαφάνεια, διότι πολύ συχνά η Κίνα έχει μία συντεχνιακή προσέγγιση ως προς τη διαχείριση αυτών των επιχειρήσεων. Ε, η Ευρώπη δεν έχει ένα ξεκάθαρο σύστημα επενδύσεων. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για αυτά τα πρότυπα ασφαλείας. Γιατί δηλαδή στις τηλεπικοινωνίες οι Κινέζοι ε, μπλοκάρονται ως προς τις αγορές της ΗΠΑ, αλλά όχι ως προς αγορές εδώ στην Ευρώπη. Δηλαδή εμείς είμαστε πιο ανοιχτοί και δεν ε, θέτουμε ζητήματα επενδυτικής ασφάλειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε προστατευτικοί, αλλά είναι ένα θέμα που οφείλουμε να θίξουμε. Έχω υπερβεί το χρόνο μου, γι' αυτό θα σταματήσω εδώ. Φτάσατε στα συμπεράσματα που θέλετε. Μου, μου δίνετε ένα λεπτό. 15 δευτερόλεπτα. Ως προς τις δημόσιες αγορές, Ε, θα ήθελα να πω ότι η Ευρώπη χρησιμοποιεί αυτό ε, το επιχείρημα σε σχέση με τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που μπαίνουν στην Ευρώπη. Ε, υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση που έχει προωθήσει τις δραστηριότητες της στην Πολωνία για έργα υποδομών στις οδικές μεταφορές, αλλά δεν υπάρχει μια συμφωνία δημοσίων προμηθειών, ένα GPA γενικότερο που να αφορά την προσβασιμότητα στις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει ενότητα μεταξύ κρατών μελών. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ πιο εύκολες. Νομίζω ότι η Ευρώπη θα έχει μεγαλύτερη δύναμη ως συλλογική δύναμη. Σας ευχαριστώ. Now we have, um, Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Αντουάν Μπρουνέ, πρόεδρος ε, της ΑΜΠΕ ε, το Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο, καθώς επίσης και για την πρόσκλησή σας να συστηθώ. Εγώ έχω μια μακρά καριέρα στα διοδρομία στην Κρετή Ηλιονέσε, σε ΕΦΣΕ, σε στις τράπεζες αυτές για τις αγορές και στα πλαίσια ε, αυτά ε, έχω διαπιστώσει ότι το εξωτερικό εμπόριο ήταν ε, μείζον παράμετρος για την υγεία, ε, το στένος της κάθε οικονομίας. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ εγώ στην αποσταθεροποίηση του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κίνα που οδήγησε στην αποσταθεροποίηση των δημοσιονομικών μας που όπως γνωρίζετε από τον Οκτώβριο του 2009 γνωρίζουμε αυτό το πρόβλημα με το ελληνικό χρέος ε, λοιπά. Ε, εγώ πώς ε, ποια ανάγνωση έχω από τους πελάτες μας. Από το τέλος του 2009 εξεράγει η οικονομία στην Κίνα και αυτό αποσταθεροποίησε την οικονομία και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ξαφνικά το ισοζύγιο τους των εμπορικών συναλλαγών από το 2001 και μετά κατέρευσε και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης λόγω των σχέσεων με την Κίνα. Από το 2001 υπάρξει πλήρη συσχέτιση της κατάρρευσης ε, του εμπορικού ισοζυγίου Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών αφενός και αφετέρου ε, το κολοσιαίο εμπορικό πλεόνασμα στην Κίνα. Αυτή λοιπόν η δεδομένη και αποδεδειγμένη συσχέτιση ε, πρέπει να δει τι είναι το αυγό και ποια είναι η κότα. Ε, η κότα είναι η στρατηγική μερκαντιλιστική της Κίνας που από το 2009 μπήκε, στο, ένα, μπήκε στον ΠΟΕ και ε, είναι τεράστια τα πλεονάσματα πλέον το αυγό είναι ε, το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα που υφίστανται συστηματικά και ταυτόχρονα από τα τέλη του 2001 είπα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, ε, η Ελλάδα, ε, η Γερμανία και οι κάτω χώρες έχουν θετικό ισοζύγιο διότι έχουν τα πλεονάσματά τους από τη Γαλλία και την Νότια Ευρώπη. Με την Κίνα έχουν έλλειμμα. Οι κινέζικες αρχές Ισχυρίζονται ότι όλα αυτά συνέβησαν επειδή κατέρευσε η εσωτερική ζήτηση στι ΗΠΑ και στι Ηνωμένε Ενώ στην πραγματικότητα ε, αυτό οφείλεται σε ένα ε, βίαιο σοκ ανταγωνιστικότητα, βίαιο σοκ εξωτερικού εμπορίου που του ε, επέβαλε η Κίνα από το 2001 και από τη στιγμή που κατάφερε να προσχωρήσει στον ΠΟΕ. Ακριβώς εκείνη την εποχή, τέλη του 2001, ε, ήταν θωρακισμένη με ωραίο κόστος ε, τεράστιας ε, ανταγωνιστικότητας πάρα πολύ χαμηλό και σημαντικά χαμηλότερο από την Ευρώπη και ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2004 συνήθισα μία πολυεθνική που έλεγε ότι στην Κίνα το κόστος ήταν 80 ε, φορές μικρότερο από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Η ίδια εταιρεία, τα ίδια εργοστάσια ήταν 80 ε, ε, φορές περισσότερο το κόστος στις Ηνωμένε Πολιτείε σε σχέση με την Κίνα. Ουδέποτε έχει φανεί αυτό στη σύγχρονη ιστορία μεταξύ μεγάλων κρατών. Είναι πάρα πολύ αποσταθεροποιητικός παράγων αυτός και θα πρέπει οπωσδήποτε να το έχουμε υπόψη μας. Επιπλέον, ε, αν χρειάζεται καν ε, απόδειξη, ύφεση από τα τέλη του 2007 και στην Αμερική και στην Ευρώπη χωρίς να έχουμε βγει ουσιαστικά. Κανονικά μια τέτοια ύφεση θα ε, οδηγούσε σε ε, επανόρθωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο διότι η Κίνα εξακολουθεί να ε, καταλαμβάνει διεθνώς μερίδια της αγοράς εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης και η αυξανόμενη αυτή παρουσία της Κίνας οδηγεί στο ότι έχει ε, μείωση ε, του πλεονάσματος ε, το διατηρεί από το 2007 σταθερό, το εμπορικό της πλεονάσμα. Σε σχέση λοιπόν με αυτή την κατάσταση, είτε πρόκειται για τις ΗΠΑ είτε για την, Κίνα, για την Ευρώπη, συγγνώμη, υιοθέτησαν συγκυριακές πολιτικές αντισταθμιστικές. Για ποιο λόγο, γιατί κάποιος που έχει τόσο σημαντικό και συνεχιζόμενο ε, έλλειμμα στο ισοζύγιο βλέπει για το ε, εισόδημά του να μειώνεται και ε, δεν μπορεί να απορροφά ε, και μόνο από την εσωτερική του ζήτηση ε, την παραγωγή του. Άρα δεν υπάρχει ανάπτυξη, αμφισβητείται η ανάπτυξη και η διαδικασία της και ε, αποστοθεροποιείται πάρα πολύ έντονα. Γι' αυτό το λόγο διαπιστώσαμε και στι Ηνωμένε Πολιτείε και σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε από το 2001 στο 2007 αντισταθμιστικέ πολιτικέ ανάλογα με τη συγκυρία δύο ειδών. Πρώτον, μεγάλε κατηγορίε, η οικοδομή και το δεύτερο ε, ε, ε, αύξηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού. Ξέρετε ότι στις χώρες που στράφηκαν προς τις κατασκευές για να ε, ξεφύγουν προς τα εμπρός. Καταλαβαίνετε και γνωρίζετε ότι πρόκειται για τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και για δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Και οι τρεις αυτές χώρες λοιπόν, είπα ε, Βρετανία και ε, Ισπανία έδωσαν το βάρος στις κατασκευές ε, κατοικίας. Ο δεύτερος είναι το έλλειμμα του προπολογισμού και εκεί αναγνωρίζονται χώρες όπως είναι η Γαλλία, η ε, Ιταλία, το Βέλγιο, Πορτογαλία και η Ελλάδα από το 2001 στο 2007 άφησαν ε, το έλλειμμα του προπολογισμού να διονγκωθεί αλλιώς θα είχαν γνωρίσει ύφεση ακόμα πριν το 2007. Το πρόβλημα λοιπόν, καταλαβαίνετε που το πάω, είναι ότι αυτέ οι δύο αντισταθμιστικέ πολιτικέ με βάση τη συγκυρία είναι μεν ε, αποτελεσματικές βραχυπρόθεσμα αλλά δεν μπορούν να απαγιωθούν διότι βρίσκουν τα όρια τους κάποια στιγμή και από εκεί και πέρα είναι δύσκολο να ε, ασκηθεί η ίδια αντισταθμιστική πολιτική. Σε ό,τι αφορά τι χώρε που στράφηκαν προ την οικοδομή το πρόβλημα του τώρα είναι ότι όταν τα νοικοκυριά που είχαν αρχικά τη δυνατότητα να αγοράσουν κατοικία με στεγαστικό δάνειο ε, κατέρευσαν ε, ή ε, εξαντλήθηκαν, οι μόνοι οι φυστάμενοι αγοραστές δεν ήταν φερέγγι, εξού και η ιστορία των subprime και έτσι κατέρευσε η αγορά της οικοδομής στραγγαλίστηκε, πνίγηκε και ακολούθησε βαριά κρίση στην οικοδομή και τελικά στις τράπεζες και χρειάστηκε κρατική επέμβαση για να είναι δανειστής τελευταίας καταφυγής των τραπεζών με αύξηση σημαντική τότε του ε, δημοσίου χρέους. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δεύτερη μέθοδο, δηλαδή ε, να αφήσεις να σου ξεφύγει το έλλειμμα του προπολογισμού, γνωρίζετε καλύτερα από μένα τι σημαίνει. Euh, Μια χώρα που επιλέγει να διατηρήσει την ανάπτυξή της με δανεισμό εκτίθεται ε, σε τεράστια αύξηση του δημοσίου χρέους χρόνο με το χρόνο μέχρι που ε, οι πιστωτές αρνούνται γιατί ανησυχούν ιδιαίτερα οι ε, ξένοι ε, και ανησυχούν για τη δυνατότητα της χώρας να εξυπηρετήσει ε, το χρέος ε, και τις προθεσμίες και όταν αρχίζουν να ανησυχούν οι πιστωτές έχουμε αρχή δημοσίου χρέους. Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα τέλη του 2009 και τώρα συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προτιμώ να μην τις αναφέρω. Euh, Βλέπετε λοιπόν ότι η στρατηγική της Κίνας που συνίσταται στο να στοχεύει και να επιτυγχάνει τεράστια εμπορικά ε, πλεονάσματα σε σχέση με άλλες χώρες και κυρίως στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ αποσταθεροποιητική. Γιατί τώρα που βρισκόμαστε ε, το φθινόπωρο του 2011 δεν μπορεί ε, κανείς να στραφεί πλέον στην οικοδομή για να έχει μια αξιοπρεπή ανάπτυξη ούτε στην Αμερική ούτε στην Ευρώπη και ούτε το δημόσιο χρέος μπορούμε να επιβαρύνουμε γιατί υπό την πίεση των πιστωτών οι χώρες που είχαν να μπει σε αυτή την ατραπό τώρα ε, αναγκάζονται ε, βιαίως να ανακρούσουν πρίμνα. Λοιπόν, είναι συστημική αυτή η αποσταθεροποίηση πλέον και οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι χώρες της Ευρώπης υφίστανται το δηλητήριο των τεραστίων ε, ε, εμπορικών λιμάτων σε σχέση με την Κίνα και δεν μπορούν και να τα αντισταθμίσουν με τον τρόπο που έπραταν ε, και με ευφύ τρόπο μέχρι στιγμή. συμπέρασμα. Έχει έρθει η ώρα οι ευρωπαϊκές χώρες να συνέλθουν, να αντιδράσουν και να τροποποιήσουν σημαντικά την πολιτική ε, της Κίνας στο Αμερικανικό Κογκρέσο, τουλάχιστον στη Γερουσία, ξέρετε ότι αυτό τον καιρό ε, ζητούν ε, να αλλάξει η ισοτιμία του νομίσματος. Αν ακολουθήσει αυτή τη γραμμή η, Αμερική θα ήταν κρίμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μείνει εκτός ιδιαίτερα όταν η ΗΠΑ συμμαχίσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισοτιμία του Ιωάν, έχουμε πιθανότητες να επιτύχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Τζόναθαν Χόλσλαχ, ο οποίος είναι επικεφαλής τμήματος έρευνας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βρυξελών Συνικών Μελετών στην στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου απευθύνατε την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση. Υπάρχει μία παρουσίαση στην οθόνη. Όπως βλέπετε στον τίτλο, έχω βγάλει το ερωτηματικό που ήταν στην ε, πρόταση αυτή. Ε, το κυριότερο σημείο εδώ είναι ότι θα πρέπει να δούμε αυτή την ανισομέρεια από την προοπτική και να δούμε ποια είναι η ευθύνη για την επανόρθωση αυτού του ισοζυγίου, αυτής της ισορροπίας. Είναι μια κοινή ευθύνη. Θα θέλω να δω πρώτα απ' όλα την Κίνα ως ένα εμπορικό ανταγωνιστή. Θέλω να δω πόσο ε, πόση ανταγωνιστικότητα κερδίζει η Κίνα. Δεύτερον, κάποια στατιστικά στοιχεία για την, ε, το σύμμετρο εμπόριο. Επίσης, κοινή ευθύνη και αν έχουμε χρόνο μπορούμε να αναπτύξουμε ορισμένα σενάρια. Έχουμε ετοιμάσει μια μελέτη σχετικά με τις συμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και την Ευρώπη, όπου βρήκαμε ότι η συμπληρωματικότητα η εμπορική που συγκρίνει όλες τις εξαγωγές με λεπτομερή τρόπο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα, η συμπληρωματικότητα λοιπόν έχει μειωθεί κατά 20% τα τελευταία 10 χρόνια, που σημαίνει ότι οι Ευρωπαϊκέ εταιρείε τώρα έχουν 20% ε, μεγαλύτερο ανταγωνισμό από την Κίνα και η Κίνα έχει γίνει ανταγωνιστής γενικά σε 36% των αγαθών που εξάγουμε. Αυτό ε, δεν ε, είναι στο βαθμό που έχουμε την επικάλυψη ε, με, άλλες, με άλλους εμπορικούς εταίρους όπως η ΕΕΠΑ και άρα ε, θέτουμε, ε, βλέπουμε από κάποια προοπτική την ανταγωνιστικότητα της ε, Κίνας. Η συμπληρωματικότητα θα μειωθεί διότι βλέπουμε την Κίνα να μπαίνει σε στρατηγικές βιομηχανίες φαρμακευτική, στην βιομηχανία, στην αεροναυπηγική. Εάν η Κίνα θα υλοποιήσει τα σχέδια για αυτές τις βιομηχανίες, αυτό θα σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό, όχι μόνο σε διμερές εμπόριο, αλλά και ανταγωνισμό από τρίτε αγορέ. Επίσης, ένα σημαντικό έβριμα τη έκθεση που θα εκδοθεί σε μερικές εβδομάδες είναι ότι μόνο ένα μικρό μερίδιο ε, του ε, συγκριτικού πλεονεκτήματος ε, της Κίνας οφείλεται σε κυβερνητικέ παρεμβάσει. Μόνο 13% οφείλεται στις τρευλώσεις των κεφαλαίων, στα φτηνά δάνεια, το γεγονός ότι η Κίνα έχει ε, χαμηλότερα εργατικά, έχει όμως καλύτερη ε, υποδομή, ε, σταθερό πολιτικό περιβάλλον, αυτό κάνει τη διαφορά. Δεύτερο σημείο, ανισομερές εμπόριο. Δεν βλέπω ε, να βιάζονται να μπουν στην Ευρώπη. Βλέπω ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες περισσότερο θέλουν να πάνε στην Κίνα ε, και αυτός ο πίνακας δείχνει τις καθαρές εκροές στο ισοζύγιο πληρωμών και τις καθαρές εισρωές και καθιστά σαφές ότι πρέπει να πάμε πέραν από το εμπόριο των αγαθών και των υπηρεσιών, αλλά έχουμε και κάποιες σημαντικές καθαρές έκροες ή ελλείμματα σε ό,τι αφορά τις άμεσες επενδύσεις, άλλες επενδύσεις που καλύπτουν πολλές ε, εξαγωγές και επίσης στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, στις τρέχουσες μεταβιβάσεις ε, και ε, αυτό είναι σε αυτό οφείλεται η ανισομέρεια στις εμπορικές ε, σχέσεις μας. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι ε, κατά πόσο η Κίνα ε, αντισταθμίζει το έλλειμμα ε, με τις αγορές αποθεματικών στοιχείων ενεργητικού. Ε, δεν έχουμε επίσημα στατιστικά στοιχεία, αλλά υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή κάπου 450 ως 550 των ε, στοιχείων ενεργητικών έχουν αγοραστεί από την Κίνα, που είναι καλό. Όχι τόσο σε βαθμό ε, που αγοράζουν οι ΥΠΑ, αλλά είναι σημαντικό ο βαθμός. Γενικά ε, τα τελευταία πέντε χρόνια είχαμε σορευμένο έλλειμμα ή εκροές στο ισοζύγιο πληρωμών 500 δις δολαρίων είπα Φαίνεται πολύ ε, ανησυχητικός ο αριθμός, αλλά αντιπροσωπεύει μόνο το 0,3% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Άρα είναι μια καλή, ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί ε, μπορούμε να εξωτερικεύσουμε ε, πολλές από τις βιομηχανικές δραστηριότητες που ίσως να μην θέλουμε να έχουμε εδώ πια. Γενικά ε, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας είναι δραματικό αλλά γενικά δεν πρέπει να το βλέπουμε έξω από τις διαστάσεις του και δείχνει επίσης ότι η Κίνα δεν είναι από μόνη της υπεύθυνη για τις ασύμετρες εμπορικές σχέσεις που έχουμε με την Κίνα. Υπ' αυτή την έννοια ε, υπήρχαν διπλές στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και, όλα και δεν είναι όλα αποτέλεσμα του κινέζικου ε, μερκαντιλισμού. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και το έλλειμμα περνάει τώρα από τις ασιατικές χώρες στην Κίνα. Θέλω τώρα πολύ διαστικά να δούμε αυτή την διπλή ε, διτή ε, στρέβλωση γιατί ο συνάδελφος έχει ήδη αναπτύξει το θέμα στην προηγούμενη παρουσίαση αλλά ε, το ασύμετρο εμπόριο με την Κίνα δείχνει ότι έχουμε αναπτύξει δύο διαφορετικές μοντέλα οικονομικής μεγέθυνσης που έχουν φτάσει στα όρια τους. Στην Ευρώπη έχουμε ε, μια κατανάλωση που οθείται από το έλλειμμα, ενώ στην Κίνα είναι μια αύξηση που ε, οθείται από το πλεόνασμα. Έχουμε ε, έχουμε φτάσει στα όρια και στην Ευρώπη είχαμε τις, την κρίση που ήταν αποτέλεσμα της κατάστασης. Αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή η διπλή στρέβλωση που ουσιαστικά και αναπόφευκτα χρειάζεται μια διπλή ρύθμιση. Δεν πρέπει να αναμένουμε μόνο από την Κίνα από μόνη της να εξυγχρονιστεί, να αυλευθερωποιήσει την οικονομία της. Το πρέπει να αντισταθμίζεται από σοβαρές ε, ε, ε, επανορθώσεις και στην Ευρώπη και θα πρέπει να υπάρχει μια αποφασιστική εμπορική πολιτική Ποια είναι τα σενάρια. Υπάρχουν πέντε διαφορετικά σενάρια τα οποία θα μπορούσαμε να εξετάσουμε. Πρώτα, να αφήσουμε τις αγορές να δουλέψουν από μόνες τους και να ρυθμιστεί η κατάσταση από τις αγορές. Νομίζω δεν έχουμε ε, πολύ χώρο να κινηθούμε εδώ. Δεύτερον, να προχωρήσουμε όπως είναι τα πράγματα και η Ευρώπη να υιοθετήσει το μοντέλο της ΕΠΑ, δηλαδή να καλέσουμε ε, τους Κινέζους να αγοράσουν περισσότερα στοιχεία του ενεργητικού ε, για να διατηρήσουμε τα βιωτικά επίπεδα, γιατί ε, αλλά δεν ξέρω αν οι Κινέζοι ενδιαφέρονται να το κάνουν αυτό, δεν θα δουλέψει. Τρίτον, υπάρχει ο προστατευτισμός και η εμπορική πόλεμη που έχουμε έχουμε ε, χρησιμοποιήσει για να κλείσουμε μέρη των δικών μας αγορών. Δεν νομίζω να οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερο σενάριο, τέταρτο σενάριο, ε, σταθερή συντονισμένη ρύθμιση που θα δει μια εξασθένηση του ευρώ. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε κάποιο πλέον έκτημα σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές και μια ενίσχυση του UN, ε, και ε, θα πρέπει να... Ε, και ούτε και αυτό δεν θα συμβεί. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι δεν είναι και τόσο ακαδημαϊκή αυτή η αξιολόγηση. Είναι ότι θα πρέπει να πάμε στο πέμπτο σενάριο που είναι βραχυπρόθεσμα να προσποιούμαστε ότι ακόμα συνομιλούμε και ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση ε, στην ασυμμετρία και τα στρες που υπάρχουν και τις εντάσεις, αλλά αυτό δεν θα βοηθήσει πάρα πολύ ε, στο να επανορθώσει τις ανισομέρειες που, ε, που είναι υποκείμενες και θα οδηγήσει σε περισσότερη αστάθεια και πανικό μακροπρόθεσμα και σε τελευταία ανάλυση πιστεύω θα αυξήσει τον προστατευτισμό και από τις δύο πλευρές, όχι μόνο από την πλευρά της Ευρώπης, αλλά αυτό είναι πιθανό να συμβεί και στην Κίνα και η Κίνα μπορεί τελικά να κλείσει κάποια μέρη της οικονομίας της περισσότερο από ό,τι σήμερα οι συστάσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρώτον, να μεταφέρουμε την προσοχή στην Κίνα. Αυτό θα μπορούσε να ήταν θετικό πολιτικό, αλλά οικονομικός είναι επιβλαβέ. Η κυριότερη λύση ε, στο ασύμετρο εμπόριο είναι να λύσουμε τις ε, εσωτερικές ανισορροπίες μας. Ε, να ζητήσουμε και να φέρουμε την Κίνα να ανταποδώσει στις εσωτερικές μας μεταρρυθμίσεις. Και τελικά ε, να δούμε, να λύσουμε τη δική μας οικονομική, ε, τα οικονομικά προβλήματα και να τιμωρήσουμε, να επιβάλλουμε κυρώσεις στην Κίνα εάν υποσκάπτει τις δικές μας μεταρρυθμίσεις. Με αυτά θα ήθελα να κλείσω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δέκα λεπτά ακριβώς. Mr. Viorel Bodure ο κύριος Βιωρέλ Ιστιτσόα Μπουντούρα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις ε, σχέσεις με την ε, Νοτιοανατολική Ασία και σχέσεις με την Ασία γενικότερα. Διευθύνων Σύμβουλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι ο Σάιμος Γκαλέσπη, ο διευθυντής που ασχολείται με θέματα ε, Ασίας, ο κύριος δεν μπόρεσε να έρθει εδώ. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω γιατί καλέσατε την ΕΕΔ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ελπίζω να συνεχιστούν αυτές οι συναντήσεις και στο μέλλον. Το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι οικονομικές πιέσεις ανά τον κόσμο και βεβαίως οι εμπορικές συναλλαγές. Όπως ξέρετε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητηθεί και μετά θα έχουμε την 14η διάσκεψη Ευρώπης ε, και στη συνέχεια τη συνάντηση των G20 στις Κάνες. Δεν χρειάζεται να σταθώ στο γεγονός ότι η Κίνα είναι ένας μεγάλος ε, εμπορικός και οικονομικός παίκτη. Είναι πολύ σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση Μιλήσαμε για τις διμερείς σχέσεις, αλλά όπως είπε και ένας ομιλητής, η εικόνα είναι πιο περίπλοκη γιατί η Κίνα έχει μεγάλη ζήτηση πρώτων υλών, ιδιαίτερα από την Αυστραλία και τη Βραζιλία. Επίσης αυξάνονται οι τιμές των πρώτων υλών και αυτό σημαίνει ότι οι δικές μας βιομηχανίες θα πρέπει να προσαρμοστούν οικονομικά. Επίσης έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της ανταγωνιστικότητας των κινέζικων προϊόντων. Υπάρχει μεγάλη λοιπόν πίεση προς την ε, Καμπότζη, το Βιετνάμ, την κλωστοϊφαντουργία να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. Ως προς τελευταία παρουσίαση δεν έχει νόημα να μιλάμε για διμερές πλεόνασμα αλλά για το συνολικό πλεόνασμα που απέκτησε η Κίνα. Και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι απόρριες αυτής της κατάστασης. Η κατάσταση δεν είναι η ίδια με την πρόκληση που αντιμετωπίσαμε με την Ιαπωνία τη δεκαετία του 70 με 80. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια χώρα που αναπτύσσεται με τάχιστους ρυθμούς. Η Κίνα επίσης αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε μια στρατηγική οικονομική εταιρική σχέση για να αντιμετωπίσουμε και τις κλιματικές αλλαγές καθώς και, την, και τις χρηματοοικονομικές πιέσεις. Παράλληλα θέλουμε ε, έμπρακτα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις εμπορικές συναλλαγές και τις οικονομικές συναλλαγές έτσι ώστε να έχουμε κάποιο κέρδος. Και σε προγενέστερες διασκέψεις αντιμετωπίσαμε παρόμοια θέματα και στην τελευταία θα θέλαμε να παγιοποιήσουμε μια κατάσταση, να αναγνωρίσουμε δηλαδή τρόπους συνεργασίας με την Κίνα θετικά έγινε λόγος για το Εθνικό Οικονομικό Πρόγραμμα της Κίνας και τις οδούς που διανοίγει για μας. Εμείς θα θέλαμε επίσης η Κίνα να συνεργαστεί περισσότερο με μας σε διεθνή ζητήματα. Θεωρούμε ότι μπορεί να επιτύχει περισσότερα για να προωθήσει τη σταθερότητα στο Μιανμάρ, στο Αφγανιστάν και στο Ιράν. Θα θέλαμε λοιπόν η Κίνα να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση ως παράγον σταθεροποίησης. Θα θέλαμε όμως να την πείσουμε να συνεργαστεί μαζί μας σε θέματα παγκοσμίων προκλήσεων, όχι μόνο σε επίπεδο G20. Μας ενδιαφέρει η πρόσβαση στην αγορά, θέματα αγοράς και εμπορίου και βεβαίως μας απασχολούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Προσπαθούμε λοιπόν να προχωρήσουμε με βάση αυτή την ατζέντα, με βάση ένα στρατηγικό στόχο και έναν έμπρακτο εμπορικό στόχο. Μιλάμε λοιπόν για μία συντονισμένη προσέγγιση, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διάσκεψη έτσι ώστε να πείσουμε την Κίνα να βρεθεί στο προσκήνιο των G20 και να εκφραστεί ελεύθερα. Το θέμα είναι επίγον. Δεν μιλάμε να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσει ανταλλάγματα. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ θα έχουμε χαμηλότερη ζήτηση, εγχώρια ζήτηση. Αυτό σημαίνει χαμηλότερη ζήτηση στις εξαγωγές και από αυτό θα πληγεί η Κίνα. Άρα ίσως η κινέζικη οικονομία να μην έχει τους ίδιους ρυθμούς που είχε δύο χρόνια πριν. Άρα δεν θα μπορέσουν να γίνουν πολλές επενδύσεις σε έργα υποδομής. Γι' αυτό και η Κίνα θα πρέπει να προβάλλει ξεκάθαρα τη στάση της στο G20 και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τους Κινέζους ηθήνοντες να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλάμε για, τα, για καλύτερα δίκτυα πρόνοιας, υπάρχει και το θέμα του νομίσματος, υπάρχουν χρηματοοικονομικά θέματα γενικότερα. Όλα αυτά τα θέματα θα τα θίξουμε στη διάσκεψη. Ελπίζουμε οι Κινέζοι να είναι πιο θαραλέοι Αν δεν έχουμε θετική έκβαση από το G20, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Μπορεί να συμβεί, αλλά δεν θα ήταν καθόλου θετικό για μας. Πολλοί μίλησαν για έναν κατακαιρματισμό προσέγγισης, αλλά ήμουν παρόν στο Συμβούλιο ε, Υπουργών Εξωτερικών χτες και ε, έχουμε σαφείς απόψεις για το τι θα πρέπει να επιδιώξουμε από αυτή τη διάσκεψη ε, κορυφής με την Κίνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος, η κυρία Έλενα Κένιχ της ε, Επιτροπής από την Γενική Διεύθυνση Τρεν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή σας καθώς επίσης και τη γραμματεία. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να συμμετέχουμε και να σας βοηθήσουμε για την προετοιμασία των συζητήσεων και της έκθεσής σας. Βέβαια, το θέμα της Κίνας είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε στα θέματα του εμπορίου σήμερα και είναι ενδιαφέρον ακούγοντας απόψεις παντού στην Ευρώπη, όπως και εδώ σήμερα, συμφωνούν όλοι για το ποιες είναι οι προκλήσεις και πόσο μεγάλες και ευρείες είναι. Είναι γεγονός ότι η Ασία και η Κίνα προκειμένου είναι η ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και πολλές από τις απόψεις που εκφράστηκαν σήμερα είναι αντίστοιχες εκείνων που λέει το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο ε, στην Κίνα. Ε, ανέφεραν κάποια στοιχεία, ακούσαμε και σήμερα, για τα κέρδη των εταιριών, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι. Είναι δύσκολο για ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κίνα βεβαίως είναι μεγάλη πηγή των ιδίων τους κερδών. Και η ίδια η κινέζικη αγορά ε, τους δίνει κέρδη. σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 37% πέρυσι. Βέβαια, αυξήθηκαν με μικρότερους ε, ρυθμούς από ό,τι οι εισαγωγές μας. Κυριαρχεί η χαλιβουργία στις εξαγωγές ε, είναι από τις μεγαλύτερες αγορές και τις μεγαλύτερες δυνατότητες και ελπιδοφόρες για το μέλλον. Από την άλλη όμως έχουν όλο και περισσότερο την αίσθηση και οι εταιρείε και εντός και εκτός της Κίνας ότι δεν ανοίγει τις αγορές της ικανοποιητικά η Κίνα και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι μέλη γενέστε. Είναι λίγο ε, χαρτογράφητα ύδατα Και επίσης ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ζητήματα ε, κάθε είδους που απασχολούν και προβληματίζουν και ανησυχούν ε, τις εταιρείες. Είναι η συμμόρφωση με τον ΠΟΕ, ο ανταγωνισμός, η πρόσβαση στην αγορά, πρόσβαση στις πρώτες ύλες και για τις παγκόσμιες αγορές μιλώ εδώ και για τις τιμές που ανέφεραν οι προηγούμενοι, ο προλαλής σας, αλλά και η πρόσβαση ε, στις πρώτες ύλες στην ίδια τη χώρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς κλάδους της βιομηχανίας. Και βεβαίω σας μην λησμονούμε τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και αντίκτυπο, πολύ δε περισσότερο σήμερα που η Κίνα ε, δαπανά πάρα πολύ και επενδύει στην καινοτομία έχει καταστεί αυτό πολύ σημαντικό για πολλές καινοτόμες ιδέες και υπάρχουν επιθυμίες και από πλευράς ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιριών να μπουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί εκεί αναπτύσσεται η αγορά. Επιτρέψτε μου να μπω σε λεπτομέρειες μερικά από αυτά τα ζητήματα. Εμείς ε, επιμένουμε πάρα πολύ στο διάλογο που έχουμε με τους Κινέζους για αυτά τα θέματα και εγώ επί σειρά ετών τα παρακολουθώ. Επιτρέψτε μου να αναφέρω πρώτα ίσως τα θετικά. Βέβαια, έχει και αυτό δυσκολίες και προκλήσεις. Το είπαν και κάποιοι προλαλήσαντε ότι βολιδοσκοπούμε τις δυνατότητες υπογραφής μιας επενδυτικής συμφωνίας. Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση, αλλά και η ευρωπαϊκή πλευρά και η κινέζικη πλευρά έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, το παρακολουθούν, το μελετούν και είναι εύκολο θα έλεγε κανείς να δούμε τις δυνατότητες και στις δύο πλευρές προστασία των επενδύσεων είχαμε περισσότερο εμείς, ε, αλλά τώρα που έχουμε δυνατότητα κοινή αντιμετώπισης Λοιπόν, η προστασία των επενδύσεων ενδιαφέρει περισσότερο τους Κινέζους και τους Ευρωπαίους η πρόσβαση στις αγορές η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ περισσότερες ε, κινέζικες επενδύσεις από ότι αντίστροφα. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κατάλογο επενδύσεων που χρησιμοποιούν για να καθοδηγούν πού χρειάζονται και θέλουν επενδύσεις, αλλά και όταν πρόκειται για θέματα προτίμηση εταίρου, κοινοπραξίες, ε, ανώτατο όριο ροφή στις ε, μετοχές και στις συμμετοχές. Αν λοιπόν μπούμε σε διαπραγματεύσει για συμφωνία επενδυτική θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι στο τέλο θα υπάρχει ένα τελικό προϊόν εντός εισαγωγικών που θα έχουμε συμφωνήσει και διαπραγματευτεί με του κινέζου και θα δίνει περισσότερε δυνατότητε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν και πιο ασφαλεί επενδύσει στην Κίνα αλλά και μεγαλύτερη πρόσβαση στην κινέζικη αγορά. Αυτό το συζητούμε τώρα με του ομολόγου μα στην Κίνα. Παραδοσιακά η ε, Κίνα δεν έχει τέτοιες ε, συμφωνίες διαπραγματευτεί που να περιέχουν διατάξεις για την πρόσβαση στην αγορά, για διάνοιξη της αγοράς τους. Θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο τελικά να συμφωνήσει η Ευρώπη σε μια επενδυτική συμφωνία που να μην περιέχει καμία ρήτρα για διάνοιξη των αγορών. Ένα άλλο τομέα που νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό για ανάπτυξη είναι ο μέσο των υπηρεσιών ε, μιλούμε εδώ για υπηρεσίες, εμπόριο έτσι και ε, μεταξύ Ευρώπης και Κίνας 16 ε, δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές από την Κίνα και 20 δις. Εκεί έχουμε 4 δις ένα ελαφρύ πλεόνασμα στις υπηρεσίες. Είναι ο δεύτερος εταίρος μας. Η πρώτη είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι 131 και 125 αντίστοιχα ε, ε, το εμπόριο στις υπηρεσίες συνολικά 250 δισεκατομμύρια. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλο έδαφος για αύξηση των υπηρεσιών με την Κίνα και οι Κινέζοι το έχουν εντοπίσει, το έχουν αντιληφθεί ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί και αγορά τους. Λοιπόν, ε, αν ε, μου επιτρέπετε να περάσω στα πιο ακαθόδη ζητήματα. Σας είπα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και βεβαίως ε, και στα νομικά ζητήματα γίνεται πρόοδος ακριβώς με την πνευματική ιδιοκτησία, αλλά έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην εφαρμογή. Εκεί πραγματικά είναι το κλειδί. Πώς θα βεβαιωθούμε ότι οι εταιρείε πραγματικά προστατεύονται με τον τρόπο που υποτίθεται ότι προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο. Είναι πολύ ε, σημαντικό αυτό και να είναι απλή η διαδικασία, να μην ε, τραβάει σε μάκρος ε, χρόνια ολόκληρα. Επιμένουμε πάρα πολύ ε, και προς τους Κινέζους ομολόγους μας και συναδέλφους ότι είναι και προς το συμφέρον της Κίνας να έχει ισχυρή προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και συμφωνεί και η Κίνα. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι και τι λέγουμε εμείς ότι βεβαίως προχωρούμε αλλά θα πρέπει και εκείνα να προχωρεί με ταχύτερους ρυθμούς, αλλιώς θα είναι εις βάρος της, της ίδιας της ανάπτυξής της. Βεβαίως και προφανώς είναι σημαντικό αυτό όταν γίνεται λόγος για την καινοτομία, όπως είπα προηγουμένως, γιατί εκεί είναι το κλειδί της ε, ε, οικονομίας και της καινοτομίας, το να είσαι κάτοχος των δικαιωμάτων. Ε, τα δημόσια έργα κρατικές προμήθειες, βεβαίως δεν είναι ε, συμβαλόμενο μέρος στη διακρατική συμφωνία η Κίνα για τις κρατικές προμήθειες, αλλά πολλά δημόσια έργα γίνονται και εμπίπτουν σε ε, άλλο νόμο. Και το θέμα είναι η πραγματική πρόσβαση στα έργα. Δεν είναι απαραίτητο όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες εκτός οποιασδήποτε σύμβασης, αλλά θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και με τρόπο διαπραγματευμένο, να ξέρουν ε, δηλαδή οι εταιρείε ότι έχουν αντίστοιχη πρόσβαση στις κοινέ αγορές όπως και οι Κινέζοι στην ευρωπαϊκή αγορά των δημοσίων έργων. Και ένα τελευταίο θέμα, αν μου επιτρέπετε, είναι ε, το θέμα των επιδοτήσεων και των ε, επιδοτήσεων των εξαγωγών το έχουμε συζητήσει και εσωτερικά. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και προσπαθούμε να αρχίσουμε ένα διάλογο με τους Κινέζους υπουργούς. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού που χειρίζεται αυτά τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων, ενώ στην Κίνα είναι κατακαιρματισμένα και διάσπαρτα αυτά τα θέματα σε διάφορες υπηρεσίες, οπότε δυσκολεύεται και ο διάλογος. Το δε κινέζικο μοντέλο είναι κάπως διαφορετικό από το ευρωπαϊκό ως προς τις κρατικές ενισχύσεις. Είναι πολλές οι επιδοτήσεις που δίνουν και διαφόρων ειδών οι κρατικές ε, παρεμβάσεις και εξαγωγικές επιδοτήσεις και πιστώσεις. Δεν είναι κακές όλες οι κρατικές ενισχύσεις, αλλά ε, θέλουμε να το συζητήσουμε μαζί τους. Πώς ε, θα έχουμε ένα καλό σύστημα και ίσους κανόνες παιχνιδιού χωρίς να καταργήσουμε τις ενισχύσεις. Σταματώ εδώ. Για μας είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα θέματα να τα συζητούμε, να συνεχίσουμε να το θέτουμε υπόψη τους και να πιέζουμε και να τονίζουμε τη σημασία τους. Είναι και προς το ίδιο συμφέρον της Κίνας και να πούμε ότι προχωρούμε μαζί προς τα εμπρός. Είναι τόσο αλληλένδετες, αλληλοεξαρτώμενες και η οικονομία μας και οι βιομηχανίες μας ε, που θα πρέπει να έχουμε και μια κοινή πορεία. Ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση. Τα μέλη της Επιτροπής μας. Ο Γιάννικ Ζαντό ε, από τους ε, Πρασίνους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρεμβαίνοντες. Ήταν άκρος ενδιαφέρουσες ε, οι εισηγήσει. Ε, δεν ε, μιλάμε μόνο για εφησυχασμό ως προς το τι συμβαίνει, ως προς τη χρηματοπιστωτική κρίση, τους Ευρωπαίους επενδυτές και ούτω καθεξής. Με την Ιαπωνία αντιμετωπίσαμε ένα σοκ ανταγωνιστικότητας, νοτομίας, αλλά δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με την Κίνα, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ρήξη μοντέλων, κοινωνικών μοντέλων, δημογραφικών και δημοκρατίας καθαρά, δημοκρατικών δομών. Και νομίζω ότι σήμερα ένας από τους λόγους των ε, ελλημάτων, του μεγάλου ελλείμματος, βασίζεται σε αυτή τη συγκρουσιακή σχέση. Την έλλειψη δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινωνική προστασία, δεν έχει προσυπογραφεί η σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να αναφωνήσουμε την αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι φέρει ευθύνε και η Ευρώπη διότι σήμερα το γεγονός ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική δεν μας επιτρέπει να εξεύρουμε μια στρατηγική, να ενταχθούμε στην παγκόσμια σκακέρα και ιδιαίτερα ε, ως προς μεγάλες χώρες όπως η Κίνα. Ποια είναι η σχέση μας δηλαδή. Εμείς πέσαμε σε μια παγίδα. Δηλαδή είχαμε πολύ πολυμερείς σχέσεις με, τη, με την Κίνα, χωρίς δηλαδή να μιλάει η Ευρώπη με μία φωνή. Αφήνουμε 10 δις εδώ, 15 εκεί και ο κάθε πρόεδρος είναι ικανοποιημένος λέγοντας ότι ε, έφτασε σε πολλές συμφωνίες παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα εμπορικό έλλειμμα της τάξης των 30 δις η G20 είναι ένα πολύ καλό ε, φόρουμ, αλλά, αλλά και ο Σαρκοζή ακόμα που προσπάθησε να δώσει μία σπίθα ελπίδας δεν τα κατάφερε, δηλαδή σε σχέση με ένα μοντέλο οικονομικό, κοινωνικό και εσωτερικής κατανάλωσης. Η ΕΕΔ λοιπόν με εκπλήστη το ότι έχει μία τόσο αισιόδοξη αντιμετώπιση του μέλλοντος ως προς τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο G20. Έχουμε να κάνουμε με ένα σημαντικό διακύβευμα. Τη στιγμή που είμαστε η πρώτη, εμπορική, η πρώτη παγκόσμια αγορά σημαίνει ότι θα πρέπει να ορίζουμε και συγκεκριμένους κανόνες. Το κάναμε με το REACH. Δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω γιατί σήμερα η Ευρώπη δεν μπορεί να το κάνει και σε άλλους τομείς τη στιγμή, δηλαδή που στον κοινωνικό τομέα, στα κλιματικά, στα ανθρώπινα δικαιώματα, σε όλους τους τομείς των πολυμερών σχέσεων, καταφέρνει κάτι τέτοιο γιατί δεν αποφασίζει να θέσει μεγαλύτερους όρους σοβαρότερους όρους στην Κίνα ως προς τους κανόνες που ισχύουν στον κοινωνικό τομέα, στον τομέα της υγείας, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πρόσβασης στις αγορές, διότι μας ε, πουλούν αμοιβαιότητα με ιδιαίτερα υψηλό τίμημα που δεν υπάρχει έγινε λόγος για δημόσιες προμήθειες ε, με την Πολωνία, σχέσεις Κίνας-Πολωνίας. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν και Ευρωπαίοι εργάτες που θα πάνε στην Κίνα να φτιάξουν οδικές αρτηρίες. Όχι. Άρα δεν υπάρχει αμοιβαιότητα. Μιλάμε για ανταλλαγές και συναλλαγές δύο υπήρων. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πράσινη οικονομία, για έλλειψη φυσικών πόρων, να υπάρχει κοινή προσέγγιση. Όμως έχουμε να κάνουμε με μία σύγκρουση προτύπων εδώ. Άρα η σχέση μας δεν θα πρέπει να είναι αμυντική ως προς την πράσινη οικονομία, ως προς την ενεργειακή λιτότητα, ως προς την έλλειψη πόρων. Θα πρέπει να έχουμε εταιρικές καινοτόμους σχέσεις και η Ευρώπη θα πρέπει να έχει το θάρρος όταν μιλάμε για πόρους, να μην μιλάμε για εκμετάλλευση πόρων στην Κίνα, αλλά και στην Αφρική και αλλού. Ευχαριστούμε τον Γιάννικ ε, Ζαντό ε, Βίνκλερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλες τις παρουσιάσεις που ήταν ε, σίγουρα ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα να εκφράσω κάπως την απογοήτευσή μου για τον τίτλο αυτής της συζήτησης και για την έκθεση που θα συνταχθεί, διότι η ανισομέρεια στο εμπόριο ανάμεσα στην ΕΕ και την Κίνα ίσως να είναι κάποιος ε, στενά που βλέπουμε το θέμα. Ε, θα πρέπει να δούμε την μεγαλύτερη εικόνα. Η ανισομέρεια στο εμπόριο είναι ένα κίνητρο ή είναι ένα επακόλουθο της ποιότητας και του περιεχομένου των διμερών σχέσεών μας. Είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την ε, κατάσταση των σχέσεων μας με την Κίνα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ε, δυναμικό, υπάρχει τεράστιο δυναμικό, αλλά βλέπουμε ε, και τους περιορισμούς που υπάρχουν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα που δεν πρέπει να τα παραβλέπουν οι πλευρές μας το σημαντικό, είναι από τα σημαντικά θέματα, θα μπορούσε να οριστεί ως η, ο μη ικανοποιητικός βαθμός διμερών γνώσεων και κατανόησης. Εμείς καταλαβαίνουμε ε, την Κίνα και η Κίνα κατανοεί ακριβώς ε, τι σημαίνει η Ευρώπη. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό. Έχουν γίνει κάποιοι παραλληλισμοί ανάμεσα ε, το, τα, ε, τα, το πενταετές και δωδεκαετές σχέδιο ε, της Κίνας και την στρατηγική 2020 της Ευρώπης. Δεν είναι ψευδείς παραλληλισμοί. Χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις, τις ίδιες, τις ίδιες εκφράσεις όταν φτιάχνουμε τις προτάσεις. Αλλά εδώ σταματάν οι παραλληλισμοί. Είναι απλά οι ίδιες λέξεις αλλά που δεν έχουν το ίδιο νόημα, την ίδια ερμηνεία. Σαν αντίστοιχα κείμενα δεν ορίζουν τους ίδιους στόχους. Άρα πρέπει να υπάρχει καλύτερη κατανόηση, καλύτερη γνώση ε, και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αυξηθεί ο βαθμός της αμοιβαία κατανόησης, της αλληλοκατανόησης και γνώσης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε την ε, σύμπραξη, την εταιρική σχέση και θα πρέπει να μια πραγματική στρατηγική εταιρική σχέση αν θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτή την εταιρική σχέση. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται αφελές, αλλά ε, υπάρχει κάποια δυνατότητα να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την συμπληρωματικότητα περισσότερο από τον ανταγωνισμό ε, στις ε, ε, κλιματικές αλλαγές και ε, σίγουρα ακούσαμε κάποια σενάρια. Σίγουρα θα πρέπει να αποφύγουμε τους εμπορικού ε, πολέμους και την κλιμάκωση του προστατευτισμού και θα πρέπει να αυξήσουμε την συνεργασία, πρέπει να αυξήσουμε την κοινή κατανόηση του γεγονότος ότι και η Ευρώπη και η Κίνα πρέπει πρώτα απ' όλα να επιλύσουμε τις εσωτερικές ανισομέρειες και ανισοσκέλειες και αν τις επιλύσουμε αυτές με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να λύσουμε και τις διμερείς ασυμμετρίες των εμπορικών σχέσεών μας. Για να κλείσω, νομίζω αυτό που χρειαζόμαστε είναι πιο αποτελεσματικό διμερής συντονισμό και κάνουμε καλύτερη πολυμερή συντονισμό στην ε, G20 και στο πολυμερές πλαίσιο και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ε, οδεύσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Τον Πολ Μέρφυ από την ομάδα ε, της Αριστεράς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές. Πολύ κατατοπιστικές οι παρουσιάσεις και ενημερωτικές. Έχω μια ερώτηση για την κινέζικη οικονομία που θα μπορούσατε να απαντήσετε σε σχέση με τις συνθήκες στην Κίνα. Αυτό το φαινόμενο το έχουμε δει η Κίνα αναπτύχθηκε πολύ καιρό και τα δύο-τρία τελευταία χρόνια απέφυγε την κρίση ε, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο το κράτος στην οικονομία και βλέπουμε και από τη βιβλιογραφία ότι Ε, η οικονομία στην Ευρώπη πριν την κρίση βασίστηκε σε φούσκες, ε, σε μεγάλο βαθμό στην κερδοσκοπία και, ε, και διάβασα ότι στο Σκόρδο έγινε κάτι τέτοιο, τρομερή κερδοσκοπία και τέτοια φούσκα, επίσης και στην οικοδομή. 100 40% αυξήθηκαν οι τιμές και στο Πεκίνο 800% τα τελευταία χρόνια. Και σε κάποιο βαθμό μου θυμίζει και την Ιρλανδία. Πριν από δύο-τρία χρόνια πολύ μαζική κλίμακα που είχαμε ε, τεράστια έκρηξη της οικοδομής και της στέγης με φούσκες, ο κόσμος επένδυσε με μεγάλες προσδοκίες, φούσκωσε, φούσκωσε, έσκασε, όπως και στην Ιρλανδία δηλαδή. 64 εκατομμύρια διαμερίσματα έχουν χτίσει που μένουν άδεια και αζήτητα. Και βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και το χρέος ιδιαίτερα της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Και υπάρχουν και εσωτερικές αντιφάσεις στην κινέζικη οικονομία που βγαίνουν στο προσκήνιο και μπορεί να σκάσει κάποια στιγμή αυτή η φούσκα. Ένα δεύτερο Όπως είπε και ο Γιαννίκα, αυτή η τεράστια ανισορροπία έχει να κάνει και με το μισθολογικό κόστος. Και αυτό που λέμε ε, συγκριτικό συγγνώμη, πλεονέκτημα ε, τους μισθούς Κίνας. Αυτό είναι κρίσιμο και για το κόστος παραγωγής εδώ και για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται και παράγουν στην Κίνα, αλλά και την έλλειψη ζήτηση. Τι να καταναλώσει ο εργάτης στην Κίνα που παίρνει τέτοιο μισθό. China Labor Watch λέγεται μια μη κυβερνητική οργάνωση που ψάχνει ε, να βρει την ε, αλήθεια πίσω από τα εργαστήρια αυτά, τα ηλεκτρονικά sweatshops σε τόσο χαμηλές συνθήκες ε, με υπεργολαβίες και από ευρωπαϊκές εταιρείες και δείχνει ότι γίνεται τεράστια εκμετάλλευση των εργαζομένων στην Κίνα και σε τεράστια κλίμακα με συνθήκες του 19ου αιώνα. δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς να κάνουν υπηρορίες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σκληρές οι συνθήκες και οι πολυεθνικές ε, που εδρεύουν στη ΣΥΠΑ και στην Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη εποφελούνται πάρα πολύ. Ας πούμε η Apple. Αν κάποιος πάει και αγοράσει ένα iPhone είναι 600 δολάρια. 6 ε, δολάρια και 54 παίρνει το εργαστήριο που ε, συναρμολογεί ε, αυτή τη συσκευή, το εργαστήριο έτσι, όχι ο και 360 πηγαίνουν στα υλικά. Δεν είναι μόνο οι κινέζικες επιχειρήσεις που προβαίνουν σε αυτή τη στιγμή εκμετάλλευση. Προφανώς είναι και κινέζικες, αλλά βλέπουμε τι γίνεται και με τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Είναι πάρα πολύ φτηνό το εργατικό δυναμικό και πάρα πολύ ικτρές οι συνθήκες εργασίας. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα την εισηγήτριά μας, την ε, Μαριέλ Ντεσαρνές γιατί δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους, καταρχήν την ε, γραμματεία της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, διότι τα κατάφερε πολύ καλά με τις ομάδες για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης και εκτίμησα ιδιαίτερα αυτά που μας είπαν οι εμπειρογνώμονες. Τους ευχαριστώ όλους και όλες. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο-τρία σημεία. Ο κύριος Μπρουνέ μας μίλησε για το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου και το έλλειμμα των δημοσίων οικονομικών μας. Αυτό βεβαίως είναι ανησυχητικό, άκρος ανησυχητικό, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να εξισορροπήσουμε αυτή την, αυτές τις συναλλαγές που είναι άνισες με την Κίνα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Όλοι μίλησαν για το θέμα της αμοιβαιότητας. Μιλάμε πολύ γι' αυτό. Και αν είχαμε μία φωνή σε θέματα αμοιβαιότητας, αυτό θα ήταν πολύ θετικό. Εμείς έχουμε μία πολύ πιο ανοιχτή αγορά στην Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα. Έχουμε πρόβλημα προσβασιμότητας στην αγορά της Κίνας και στις δημόσιες προμήθειες, στην Κίνα και ιδιαίτερα ως προς τις καινοτόμες αγορές, διότι οι Κινέζοι έχουν μία μακροχρόνια στρατηγική. Εδώ υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός και αποφάσεις για τα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια. Και οι τεχνολογίες εχμής παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος της τούρτας. Και αυτό αφορά και τα δικά μας διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Ως προς τις εξωτερικές επενδύσεις μιλήσαμε για τη γνώση ότι υπάρχει μεγάλος περιορισμός Γι' αυτό και η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια απάντηση ως προς τις κινέζικες επενδύσεις που θα γίνουν στην Ευρώπη στα επόμενα 5 ή 10 χρόνια. Ως προς το θέμα της πνευματικής ε, διανοητικής ιδιοκτησίας, αυτό είναι άκρο σημαντικό, γιατί αν η ε, Ευρώπη δεν κρατήσει το προβάδισμα που έχει ως προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα αύριο. Τη στιγμή που ε, κυρώνεται μια συμφωνία για τεχνολογίες εχμής θα πρέπει να υπάρχει και μεταφορά τεχνολογίας. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα υπήρχε η αντίθετη ρήτρα. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει για να δούμε τι σημαίνει έμπρακτα. Και ιδιαίτερα ως προς τη μεταφορά τεχνολογίας και την αγορά των διπλωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως προς τις πρώτες ύλες και τις σπάνιες γέες υπάρχει μία στάση της Κίνας που δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Υπάρχει και παραχάραξη ως προς την πνευματική ιδιοκτησία. Υπάρχει και το θέμα του νομίσματος γιατί δεν υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός όταν μιλάμε για το κινέζικο νόμισμα και τους κανόνες που το διέπουν. Αυτά είναι ορισμένα από τα σημεία που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα που θα ενταχθούν στην έκθεση. Έγιναν αρκετές παρεμβάσεις σε θέματα επιμερισμένης ευθύνης, κοινή ευθύνης. Θα πρέπει να επιμείνουμε για μία ε, εθελούσια πολιτική, πιο απαιτητική πολιτική από πλευράς Κίνας, τουλάχιστον εγώ θα το προσπαθήσω, και παράλληλα θα πρέπει να δούμε και τα του οίκου μας στην Ευρώπη δεν μας απαλλάσσει από τις δικές μας ευθύνες. Δεν τα καταφέρουμε καλά ως προς την πράσινη οικονομία, ως προς μια κοινή βιομηχανική πολιτική, ως προς τεχνολογίες εχμής. Άρα οι ανταλλαγές είναι άνισες, οι συναλλαγές είναι άνισες. Και όταν θέλουμε μια εξισορρόπηση σχέσεων, αν εμείς δεν διευθετήσουμε τα του οίκου μας, δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Θα ήθελα λοιπόν λοιπόν ε, να προχωρήσουμε και από τις δύο πλευρές ως προς την κινέζικη παρουσία ε, στην Ευρώπη. Ο, ο φίλος μας, ο οποίος συνέταξε αυτό το έγγραφο με τον Φρανσουά Γκοντμάν, θα πρέπει να ε, τονιστεί εδώ ότι και στις ΗΠΑ μας ενδιαφέρει, όπως και στις είπα, μας ενδιαφέρει να ξέρουμε αυτό το δημόσιο χρέος, αυτό το κρατικό χρέος, πώς επιμερίζεται. Ε, εδώ και έξι μήνες ασχολούμαι με το θέμα του δημοσίου χρέους και ήθελα να ξέρω ποιο ε, τμήμα του χρέους κατέχει η Κίνα. Κανένας δεν ήξερε να μου απαντήσει. Το ίδιο αφορά τις άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό. Δεν είναι τεράστιες, αλλά ξέρουμε ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερες τα επόμενα 5-10 χρόνια. Και όπως και είπα, θα πρέπει να διαθέτουμε ένα μέσον το οποίο με διαφάνεια θα μας ορίζει ποιοι είναι οι στρατηγικοί τομείς επενδύσεων. Αυτό κάνουν οι Αμερικανοί, θα πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Ο Γιάννικ Ζαντό έχει δίκιο ως προς το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ρεσιμότητα συναλλαγών με τήρηση ρυθμίσεων, δηλαδή τα προϊόντα ε- που φτάνουν στην Ευρώπη θα πρέπει να τηρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Να έχουμε ένα νέο πλαίσιο με προδιαγραφές στον τομέα των κοινωνικό, του περιβάλλοντος, τον οικονομικό και στα πλαίσια των πολυμερών σχέσεων. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ενωμένη Ευρώπη, ενωμένη Ευρώπη και στον τομέα των τιμών. Σήμερα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική. 27 κάνουν ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτό αφορά και τους εμπειρογνώμονες και εμάς τους βουλευτές, αλλά μην ξεχνάμε και την κοινή γνώμη διότι ένα θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη είναι οι ε, σχέσεις μας, οι εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε. Λοιπόν, τελικό στάδιο αυτής της ακρόασης. Θα ήθελα να λάβουν το λόγο οι προσκεκλημένοι μας. Η κυρία Σουκρούν έχει το λόγο για να σχολιάσει τα όσα άκουσε, αλλά έχετε περιορισμένο χρόνο. Τρία λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Κυρία Σουκρούν, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, στα γαλλικά αυτή τη φορά συμμερίζομαι τις παρατηρήσεις που έγιναν ε, από τους ε, ευρωβουλευτές και αυτό που διαπιστώσαμε κατά τη σύνταξη της έκθεσης είναι ότι δεν υπάρχει ενότητα σε ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή κλίμακα και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει μια κινέζικη βιομηχανική πολιτική που είναι σαφής, προγραμματισμένη και υπάρχει ενότητα και αυτό είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους. Επίση, συμμερίζουμε τις ε, απόψεις που έγιναν σχετικά με το, τη σύγκρουση των προτύπων. Ε, ναι, ε, το εμπόριο με την Κίνα δεν είναι το ίδιο με το εμπόριο με την Ιαπωνία κατά ε, τη δεκαετία του 70. Ε, Τώρα, ε, δεν υπάρχουν ε, τακτικές δημοσίευσεις ε, κειμένων και ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που δεν είναι διαφανές και ξεκάθαρο, αλλά έχει ελεγχθεί, αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό σημείο. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν διεθνείς κανόνες και κοινές και κανόνες στον τομέα εργασίας. Ο κύριος Παρέλο Πλέσνερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας δώσατε το λόγο. Κάποια σχόλια, ε, κάτι σχετικά με τα κράτη-μέλη και ε, δύο πράγματα που έχουμε κάνει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και όπου έχουμε κάνει μια κατηγορία ε, μια κατηγοριοποίηση ε, των σχέσεων και την επικαιροποιήσαμε πριν και μετά την κρίση και αυτό αποτελεί βάση για συζήτηση. Ευχαριστώ ε, την κυρία Σανές που έχει ακολουθήσει την πρόταση της ε, διαφάνειας. Είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σημαντικό μόνο για την Κίνα αλλά σημαντικό για τι φαίνεται να με την Κίνα να έχει μια επίπτωση, χρησιμοποιείται και στην δημόσια διπλωματία στην Κίνα δίνονται αυτές οι ψευδείς ε, ε, διασφαλίσεις. Αυτό μπορεί να έχει και επίπτωση στις ευρύτερες διμερείς σχέσεις. Κάτι άλλο σε μια από τις προηγούμενες παρουσιάσεις αναφέρθηκε το γεγονός ότι οι γενικές επιδοτήσεις δεν στρεβλώνουν σε μεγάλο βαθμό τις γυναστικές ε, τιμές και τις εξαγωγές. Είναι κάπως περίεργο. Αν ε, η Ευρώπη έχει ταυτόχρονα την ίδια ε, μελέτη, έχουμε και αντίθετα μια άλλη μελέτη που λέει ακριβώς το αντίθετο ότι έγιναν ζημιές και όχι κέρδη αν αφαιρέσουμε το κόστος της χρήσης γης και της χρήσης των, δημοσιών, των εθνικών πόρων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντων Ντουάν Μπρουνέ. Μάλιστα. Θα ήθελα να αξιοποιήσω τα λίγα λεπτά που μου δίνετε για να διαμαρτυρηθώ λίγο κατά της ιδέας ότι η Κίνα είναι η ε, της ε, παγκόσμιας οικονομίας. Το είπε νομίζω κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η είναι οι χώρες ακριβώς που υφίστανται τα εμπορικά ελλείμματα λόγω των πλεονασμάτων στις εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα, της Κίνας. Η ατμομηχανή λοιπόν είναι η και η Ευρώπη. Η Κίνα παρασιτεί στην ανάπτυξή μας. Μας στέλνει εξαγωγές πολύ περισσότερες από ό,τι εισάγει και μας επιβάλλει ε, μια πάρα πολύ χαμηλή ανάπτυξη σε εμά. Από τότε που μπήκε στον ΠΟΕ η Κίνα το 2001 έχουν υποχωρήσει οι οικονομίες των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, το G7, τη Ηνωμένης Ευρώπης. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το έλλειμμα ανανεώνεται, εδρεώνεται, παγιώνεται απέναντι στην Κίνα και είναι ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά της ανάπτυξης. Θυμάμαι Τότε που είχαμε τα ίδια προβλήματα με την Ιαπωνία λέγαμε ότι ήταν ατμομηχανή ε, της παγκόσμιας οικονομίας και εγώ από τότε διαφωνούσα. Ε, que... Το επόμενο θέμα που θέλω να σας πω είναι ότι έγινε μεγάλος λόγος για τις πολυμερείς συναλλαγές. Μα σήμερα η Κίνα είναι τόσο ισχυρή στα διεθνή φόρα που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι χρειάζεται μια συμμαχία πολύ ευρύτερη, πολύ ισχυρότερη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιταχθούμε στην Κίνα. Θυμάμαι τη Σύνοδο κορυφή της Σεούλ, Οκτώβρη-Νοέμβρη του 2010, που ήμασταν αξιοθρύνητοι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, είχαν βγει στις επάλξεις ήρθε η Γερμανία ε, να τους ε, σπάσει αυτή την προσπάθεια, να την υπονομεύσει και ε, δεν κατάφεραν να κάνουν την Κίνα να υποχωρήσει στην πολιτική των συναλλαγματικών της ισοτιμιών του Ιουάν. Θα πρέπει όλες οι χώρες του G7 λοιπόν και στο G20 να έχουν κοινή στάση και πρακτική να συμπαραταχθούν. Ευχαριστώ και τελευταίος ο κύριος Χόλσλαχ. Τέσσερα ζητήματα. Καταρχήν αυτό που είπε ο κύριος Μέρφυ κατά πόσο η Κίνα φτάνει στα όρια, στα αναπτυξιακά της όρια. Βλέπουμε ότι πραγματικά φτάνει στα όρια της, δίνονται πολλές ε, μάχες παντού και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Δεύτερον, η ανάπτυξη της Κίνας και το εμπόριο έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Βλέπουμε ότι προωθούνται οι εξαγωγές από κρατικοδίαιτους οργανισμούς και βλέπουμε ότι Υπάρχει μάλλον ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων ελέγχονται από το κράτος και αυτό αφορά και τις επενδύσεις. Επίσης, το θέμα που έθιξε ο κύριος ε, Ζαντό, κατά πόσο υπάρχει σύγκρουση προτύπων. Νομίζω ότι πρόκειται για σύγκρουση αναπτυξιακών φάσεων. Αυτό μας απασχόλησε και με την Ιαπωνία στο παρελθόν, σε σχέση δηλαδή με την διαδικασία εκβιομηχάνησης της μεταξύ των δύο μεγάλων πολέμων και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα δεδομένα θα συνεχίσουν να υπάρχουν ως προς δηλαδή με το βιομηχανικό ε, πρότυπο της Κίνας και για το μέλλον. Ως προς τις ε, πολυμερείς σχέσεις, νομίζω ότι στα πλαίσια της παγκόσμιας διακυβέρνησης οι αναπτυσσόμενες χώρες θα προβάλλουν πολύ περισσότερο τα συμφέροντά τους έναντι των αναπτυγμένων χωρών που αποτελούν μία μειονότητα και οι διεθνείς οργανώσεις που ήταν ένα μέσο υπέρ ημών θα χάσουν την, ε, τη σημασία τους. Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας σε αυτή την ιδιαίτερα ζωηρή συζήτηση και ακρόση για τις ε, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την ΕΙΕΔ που δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση και εδώ αναφέρομαι στον κύριο Περέλο Πνέστερ, Κρίν Μπρουνιέ και Χολσλαγκ. Σας ευχαριστώ όλους και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγητρία μας. Δεν τελειώσαμε. Αποχαιρετούμε τους προσκεκλημένους της ακρόασης. Το καλό να πάτε. Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, αλλά ούτε και διάλειμμα. to break. Με αναγκάζεται να κάνω διάλειμμα. Παρακαλώ όσοι εξέχεστε τις αιθούσεις, το συντομότερο και ησύχως please. Our proceedings are not yet concluded. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα, παρακαλώ. Let's allow our guests to leave the room. Ας επιτρέψουμε στους προσκεκλημένους μας να βγουν. And let's hope that the room is settled. Λοιπόν, ησυχία στην αίθουσα. Things regarding noise are improving, but not, but not. Από θόρυβο καλά τα πάμε, αλλά όχι αρκετά καλά. Καλύτερα. May I ask you to stop the Σας παρακαλώ, σταματήστε τις ιδιωτικές συζητήσεις και τα πηγαδάκια στους διαδρόμους. Έχουμε και άλλα θέματα. Thank you. Let's resume our proceedings. Items... Προχωρούμε λοιπόν στο σημείο 17. Τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου του 2009 σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστοσης για τις αγωγές βοηού κρέατους υψηλής ποιότητας από τις Ηνωμένε Πολιτείες και τον Καναδά. Είναι τμήμα μιας συμφωνίας για να τερματιστεί η κατάσταση των κυρώσεων αντιπίνων που μας είχαν επιβάλει ο Καναδάς και οι Ηνωμένε Πολιτείε λόγω ε, της διένεξης για το βόλιο κρέας με ορμόνες. Η συγκήτρια μας εδώ είναι η κυρία Γκόντελίβε Κουίσταουτ Ρόβορ. The Και της δίνω μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, βασικά δεν είναι καν νομοθετική διαδικασία αυτή η αυτόνομη ποσόστοση για τις εισαγωγέ βοηού κρέατος υψηλής ποιότητας. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η πολιτική της σημασία. Εδώ και πολύ καιρό υπάρχει μια διένεξη για το βόηο κρέας με ορμόνες και από τη μια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη είπα και ο Καναδάς. Αν δεν θυμάστε, εγώ είμαι παλιά καραβάνα εδώ και ε, χρόνια ολόκληρα αγόμαστε και φερόματος. Ε, βλέπεις, ε, ο Ρόμπερτ Στέρτη με καταλαβαίνει. Το θυμάται αυτό. Ευχαριστώ πολύ. 48.000 τόνοι είναι για αυτόνομη ποσόστοση είπα και Καναδάς και έχουν επιβάλει δασμούς. Αυτό αφορά κρέας που δεν έχει υποστεί επεξεργασία με ορμόνες. Το ζώο προφανώς, όχι το κρέας. Η δική μας απέτηση να μην δίνουμε ορμόνες ε, στα βοηδή παραμένει. Δεν έχουμε αλλάξει γνώμη. Πρόκειται λοιπόν για ένα συμβιβασμό. Βεβαίως, αυτός ο συμβιβασμός και η εφαρμογή του ε, θα έχει ε, μεγάλη συμβολική σημασία θα είναι ένα μήνυμα για τις εμπορικές συναλλαγές Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια σαφή κατάσταση και πολιτική βούληση εκατέρωθεν του Ατλαντικού και κατ' εμέ ε, θα είναι θετικό αυτό και για τις δύο πλευρές. Τα επόμενα χρόνια θεωρώ καθήκον μας και υποχρέωση να λύσουμε αυτές τις διενέξεις. Παρένθεση. Την Πέμπτη το πρωί θα συζητήσουμε και την περίφημη υπόθεση στην Ολομέλεια του Buy American. Αγοράζεται αμερικανικά προϊόντα. Λοιπόν, έχουμε πολλά τέτοια ζητήματα, περισσότερα του ενός και καλό θα είναι να τα λύσουμε. Και με τους εμπορικούς φραγμούς καλό θα ήταν να τους καταργήσουμε είναι αυτό ένα μήνυμα, έλεγα, για τη διατλαντική σχέση ως βάση της παγκόσμιας οικονομίας. Γι' αυτό το συντομότερο θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Αυτά. Είναι σχετικά σαφές ότι είμαι υπέρ αυτής της συμφωνίας. Τι άλλο να σας πω. Αλλιώς δεν θα ήμουν και εισηγήτρια, έτσι δεν είναι. Ε, εν πάση περιπτώσει είμαι υπέρ ε, της ε, συμφωνίας αυτής γιατί είμαι πεπισμένη ότι πρόκειται για καλή συμβιβαστική πρόταση εποφελεί και για τις δύο πλευρές win-win όπως το λέμε και προσβλέπω σε μια καλή και στενή συνεργασία με τους κοιόδης συγητές και τους συντάκτες και συγητές των άλλων συγγνωμοδοτουσών επιτροπών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε λοιπόν τους υπολείπους. Ε, ο κύριος Κούτας από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε και η συγγήτρια, νομίζω ότι το θέμα του βοήου κρέατος με ορμόνες ε, βλάπτει τις οικονομίες, τον ΗΠΑ, του Καναδά και της Ευρώπης με την ε, εφαρμογή κυρώσεων τύπου καρουσέλ. Φτάνουμε, θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι θα πρέπει εγκαίρως να θέσουμε σε αίσιο πέρας αυτές τις διαδικασίες. Όπως γνωρίζουμε, οι οικονομίες των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το ίμιση του παγκοσμίου ΑΕΠ και γι' αυτό οι διατλαντικές εμπορικές σχέσεις έχουν μεγάλη σημασία για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας και βλέπουμε ότι δυστυχώς επιδεινούται η κατάσταση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένες επιτυχές και θα με ενδιέφερε η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος των εμπορικών κυρώσεων και ποιες θα είναι, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος σε σχέση με την αύξηση εισαγωγών βοήου κρέατος, έτσι ώστε να μην πληγούν συγκεκριμένες περιφέρειες και κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό περιμένω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και την άποψη των συναδέλφων γιατί βρισκόμαστε σε φάση της πρωταρχικής συζήτησης. Ευχαριστώ. Thank you. Robert from e Ο κύριος Στέρντι από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ. Ε, ε, συμφωνώ σε γενικέ γραμμέ με τα όσα είπε ο κύριο Κούτα. Είναι θέμα εφαρμογή ενό μνημονίου συνεννόηση. Έχετε απόλυτο δίκιο, ε, κύριε Κούτα, ότι δεν θα έχει τέτοιε επιπτώσει ούτε για τη δική μας ε, γεωργική παραγωγή. Εγώ, ξέρετε, έχω διατελέσει πρόεδρος Επιτροπής Κτηνοτροφία ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καταλαβαίνω αυτά που λέει ο επίτροπο και το Κοινοβούλιο ε, η Επιτροπή Γεωργίας νομίζω πήγαν μαζί ε, πριν από 12 μήνες ε, στι Ηνωμένε Πολιτείε για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων συζήτησαν και σύμφωνα με τον Τόμ Βίλσακ νομίζω τον λένε τον αρμόδιο και αξιωματούχο για τη γεωργία και παρακαλώ να μου το επιβεβαιώσετε είπαν να άρουν πρότειναν τους περιορισμούς για το βόλιο κρέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει και για άλλα προϊόντα. Είναι πρόθεση του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ξέρω ότι θα το γράψει η Γκοντελίβη στην έκθεσή της, να μην εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από βοηθοί που έχουν ε, λάβει ορμόνες. Είναι θέμα ε, όχι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και θέμα εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Είναι πάρα πολύ καλό να στείλουμε ένα ε, σαφές μήνυμα και να δείξουμε καλή βούληση. Ε, ευχαριστώ. Παρακαλώ την Επιτροπή να απαντήσει σε ερωτήσεις μου. Ο κύριος Ζωζέ Μποβέ, παρακαλώ, από τους Πρασίνους. Μάλιστα. Η συζήτηση αυτή είναι σημαντική, πιστεύω, και θα πρέπει να εγγραφεί στο πλαίσιο της δεν είναι ουρανοκατέβατη. Υπήρξε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τις ορμόνες. Στη συνέχεια είδαμε τι έγινε το 1996 μετά την ίδρυση του ΠΟΕ και το πάνελ Ευρωπα... Ε, ε, είπα Καναδά Φενός και Ευρωπαϊκή Ένωση αφετέρου τη διένεξη στον ΠΟΕ. Σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε. Επίσης θα πρέπει να θεμίσουμε ένα δεύτερο στοιχείο εκτός γενικού πλαισίου τι έγινε στη συνέχεια με τις κυρώσεις επί 60 ευρωπαϊκών προϊόντων επί μία δεκαετία. Γιατί η Ευρώπη αρνείτο, ε, αρνείτο να εισάγει αυτό το κρέας. Διατηρήθηκε αυτή η άνηση και απόρριψη και πολύ καλά έκανε η Ευρώπη και είχαμε εκεί ιδιαιτερότητα στην παραγωγή. Λοιπόν, είναι σημαντικό να θυμίσουμε το πλαίσιο για να πούμε ότι σήμερα έχουμε βγει από το θέμα αυτό. Βέβαια, χρειάζεται ακόμα επιβεβαίωση και επαλήθευση των στοιχείων Αυτά που έχω εγώ είναι θετικά, να μα τα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τελευταία προϊόντα που είχαν αυτού του υπερβολικού δασμού από τι αρχέ του 2011 δεν του υφίσταται. Βέβαια θα πρέπει να μα τα εγγυηθεί όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί μια τέτοια συζήτηση γενικά για τι εισαγωγέ δεν έχει νόημα αν είμαστε ακόμα στο επίπεδο των κυρώσεων. Ε, παρακαλώ, επαλήθευση είναι, αλλά πρέπει να γίνει. Και κάτι άλλο που πρέπει να συζητήσουμε στα πλαίσια τη έκθεση αυτή είναι πώς ορίζουμε την υψηλή ποιότητα. Ποια εχνηλασιμότητα έχουμε για την υψηλή ποιότητα του βοηού και ποια είναι ε, τα μεγέθη ποια η ποσόστοση. Να μην ανοίξουμε τις θύρες τώρα για τη δεύτερη συζήτηση που θα κάνουμε σε λίγους μήνες για τις εισαγωγές κρέατος υψηλή ποιότητα, γιατί όχι, που θα προέρχεται από το Μερκοσούρ, έτσι. Προσέξτε παρακαλώ να μην μπούμε σε ένα σύστημα που ε, άρδιν και ριζικά θα αλλάξει την ε, ευρωπαϊκή παραγωγή και τη διάνοιξη των αγορών και τις εισαγωγές. Είναι ένα θέμα ισορροπίας. Uh, ο κύριος Φλάβιο Κοτούρνη από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Uh, Ευχαριστώ. Νομίζω ε, ότι πολύ σωστά οριοθετήσατε το πλαίσιο αυτής της πρότασης. Είναι κάτι το οποίο φορά τη δεκαετία του 90, τα τέλη της δεκαετίας του 90, όπου ένα πάνελ των ΙΠΑ προέβαλε το θέμα και είχαμε πολλές διαφορές επί του θέματος. Το 2009 ε, επήλθε συμφωνία με τις ΙΠΑ και στη συνέχεια και με τον Καναδά. Αυτή η συμφωνία επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κρατήσει την ε, απαγόρευση του βοήου κρέατος το οποίο έχει ορμόνες και παράλληλα να μπορεί να προβάλλει αυτή τη, αυτή τη διάταξη, αυτό δηλαδή το σχέδιο και προς τα έξω. Στη συνέχεια είχαμε έναν οδικό χάρτη για τα τρία στάδια αυτής της ε, συμφωνίας και τώρα θα φτάσουμε στη δεύτερη φάση έτσι ώστε να αρθούν οι κυρώσεις γιατί στην ουσία βρεθήκαμε πάνω από τις προσδοκίες μας και για να απαντήσω και στον κύριο Μποβέ μπορώ να σας πω ότι αυτές οι κυρώσεις έχουν αποσυρθεί και η ΕΠΑ ήραν τις κυρώσεις πριν από την απόσυρση όλη του πλαισίου που προβλεπόταν μέχρι το 2000, προβλέπεται μέχρι το 2012. Αυτές οι κυρώσεις έχουν αρθεί δηλαδή 13 μήνες πριν. Έχουν αρθεί από τη ΕΠΑ. Αυτό ήταν πολύ θετικό και το ίδιο ισχύει και με τους Καναδούς οι οποίοι ήραν όλα τα μέτρα και εφαρμόζουν τη συμφωνία, άρα οι εξαγωγές μας μπορούν να ε, στρέφονται προς τον Καναδά χωρίς επιπρόσθετους δασμούς. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο βήμα προς αυτή την ε, κατεύθυνση, δηλαδή να εφαρμόσουμε και εμείς το δικό μας σκέλος της συμφωνίας. Τα πλεονεκτήματα αφορούν όχι μόνο το εμπόριο, διότι όπως ξέρετε υπήρχε αυτή η διαφορά που είχε ολέθριες επιπτώσεις και όπως είπε και η συγγήτρια είχαν επιδεινωθεί και οι σχέσεις μας, οι εμπορικές σχέσεις με τη ΣΥΠΑ. Μετά από τη σύναψη αυτής της συμφωνίας υπάρχει θετική στάση των ΙΠΑ και σε άλλα εμπορικά ζητήματα. Δεν σημαίνει θα τα επιλύσουμε όλα, αλλά τουλάχιστον εφόσον ήραν τις κυρώσεις 13 μήνες πριν από την προθεσμία, αυτό είναι ένα σαφές δείγμα του ότι λειτουργεί καλώς αυτή η συμφωνία. Ως προς τα ιδιαίτερα ερωτήματα, δηλαδή τις επιπτώσεις του βοήου κρέατος υψηλής ποιότητας και οι επιπτώσεις των κυρώσεων, θα ήθελα να πω ότι οι κυρώσεις είχαν επιπτώσεις βεβαίως, πέρα από την ε, ποσοστοποίηση που έγινε από το Πάλεν, δηλαδή μιλάμε για 110 εκατομμύρια δολάρια. Είναι δύσκολο να ορίσουμε ποσοτικά τις επιπτώσεις των ε, κυρώσεων, διότι μιλάμε για εμπόριο και παραγωγή από τη δική μας πλευρά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επιπτώσεις σχετίζονται γενικότερα με τις εμπορικές σχέσεις, όχι μόνο με την παραγωγή βοηού κρέατος. Δηλαδή, αν δούμε τις εμπορικές και τις πολιτικές επιπτώσεις, είναι πολύ ευρύτερες. Και ήταν ουσιώδης και για τις αγορές και για τις εμπορικές σχέσεις. Αν όμως το δείτε ιδιαίτερα, ε, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλήγησαν από τις κυρώσεις και αυτό αφορά και το ε, κύριο κρέας, τα ροδάκινα, σε κονσέρβες, ροκφόρ. Και το πορτό. Και φτάσαμε και σε ένα 300, 100 με 300% αν θέλουμε να ε, θέσουμε ποσοτικούς όρους στις επιπτώσεις. Τώρα, ως προς το βόλιο κρέας, αυτό που έχει σημασία να λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για 48.000 τόνους, ε, δεν πλήττεται η αγορά βορείου κρέατος στις ΗΠΑ, ελέγχουμε την κατάσταση και εποπτεύουμε στην κατάσταση, την κατάσταση εδώ και 1,5 χρόνο όπου ε, δεν ισχύουν οι δασμολογικές ποσοστώσεις, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο όγκος των ε, δασμολογικών ποσοστώσεων και κατά πόσο μπορεί να πλήξει και να ε, κλειδωνεί στην αγορά. Ως προς σπογγόδια εγκεφαλοπάθεια, ο Επίτροπος Τσόλος έθιξε αυτό το ζήτημα πριν από το καλοκαίρι και ο κύριος Νταλή το έθιξε δύο-τρεις φορές κατά τις επισκέψεις του στη ε, Ουάσιγκτον και το θίξαμε και με τον Υφυπουργό Γεωργίας, τον είπα. Ο Υφυπουργός Βίλσεκ μας είπε ότι θα δημοσιεύσει τους κανόνες για την αντιμετώπιση της πογκόδους εγκεφαλοπάθειας των βοηδών μέχρι το τέλος του έτους. Σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει μία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με τη βιομηχανία μεταποίησης δηλαδή. Θα υπάρχουν δύο μήνες προθεσμία για να λάβουμε τα σχόλια από τους εμπλεκόμενους φορείς και μετά θα γίνει αξιολόγησή τους και στη συνέχεια θα ληφθεί μία απόφαση με βάση αυτή την αξιολόγηση. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα, δεν σημαίνει ότι θα αρθούν οι κυρώσεις άμεσα, αλλά είναι το αμέσως επόμενο βήμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κατάσταση. Έχει μεγάλη σημασία για τους εξαγωγείς μας, αλλά και για τη βιομηχανία των ΙΠΑ. Και οι παραγωγοί ε, έγραψαν στον Υφυπουργό Γεωργίας και ανέφεραν θέλουν να αρθούν αυτά τα θέματα, διότι υπάρχουν ε, σημεία τριβής μεταξύ ΙΠΑ, Κορέας και Ιαπωνίας. Γιατί θέλουν να εξάγουν στην Κορέα και στην Ιαπωνία, γι' αυτό ακριβώς οι αρχές των ΙΠΑ θα πρέπει να άρουν την απαγόρευση αυτή. Ως προς το ερώτημα του κυρίου Μποβέ, δηλαδή πώς ορίζουμε την υψηλή ποιότητα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον ορισμό του κανονισμού, ο οποίος είναι πολύ εξειδικευμένος και ισχύει για αυτό τον τύπο βοήου κρέατος και δεν μπορεί να ισχύσει γενικότερα. Δεν μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε αυτό το προηγούμενο το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο γιατί μιλάμε για έναν εξειδικευμένο ορισμό που αφορά αυτό τον τύπο βοήου κρέατος και δεν θα ισχύσει αλλού όπου θα διενεργηθούν άλλου είδους διαπραγματεύσεις. Ε, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε την Κομισιόν για αυτές τις ε, διευκρινήσεις. Λοιπόν, η συγγήτρια. Είναι πρώτη ανταλλαγή απόψεων ο πρόεδρος, ακριβώς η κυρία Κουίσταλτ. Σύντομα, νομίζω ότι γενικά συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Μερικά πράγματα χρειάζονται διευκρίνηση. Ας μην λησμονούμε ότι τελικά ε, το πάνελ στον ΠΟΕ τον χάσαμε και έκτοτε από χρόνο σε χρόνο κάνουμε διάφορα εμβαλωματικά όσα αντιδράσεις που δεν μπορούν να διονίζονται. Είναι πολύ σημαντικά μερικά στοιχεία που να επαναλάβω και εγώ. Αυτό που είπε ο κύριος Μποβέ για την ποσόστοση των Ηνωμένων Πολιτειών, να μην διαταράσσεται η ισορροπία στην ευρωπαϊκή αγορά και βέβαια και στις διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ θα ε, πρέπει να συζητήσουμε και θέματα βοήου κρέατος. Το δεύτερο, που ίσως να μην τόνισα εγώ επαρκώς, πρόκειται για κρέας από βοηδή που δεν έχουν προσλάβει ορμόνες και θα πρέπει να το τονίζουμε πάντα. Θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος των εισαγωγών. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι κόρη και εγγονή κτηνιάτρων και θεωρώ ότι γίνονται κτηνιατρικοί έλεγχοι, κρέοσκοπικοί έλεγχοι, δειγματοληπτικά και δεν ε, περιτεύουν. Καλό είναι να γίνονται και να έχουμε μία ε, διαδικασία που να μας εγγυάται ότι δεν θα συνεχίζονται οι προσφυγές, γιατί το έχουν κάνει λίγο γαϊτανάκι αυτό με τις προσφυγές στον ΠΟΕ. Το ξέρω ότι τυπικά μπορούν να το κάνουν. Σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε. Θα έρθω σε επαφή με όλους σας ξανά πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ διαφορετικά όλα αυτά που μας είπατε. Την επόμενη φορά τον Νοέμβριο στη συνεδρία της Επιτροπής θα έχουμε και το σχέδιο 22 ε, και 23 Νοεμβρίου. Ε, θα έχουμε το σχέδιο της έκθεσης. Και περνάμε τώρα στο τελευταίο θέμα, η κατάσταση ε, όσον αφορά στις προσχωρήσεις των ΠΟΕ. On my left, uh, εδώ εξεβονίμων κάθεται ο κύριος Μπάλας, ο οποίος είναι επικεφαλής διαπραγματευτής και αναπληρωτής ε, γενικός διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται ενώπιόν μας. Θα μας κάνει μια εισαγωγή. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. για να ε, ε, δούμε ποιες είναι εκτιμήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις προσχωρήσεις των ΠΟΕ. Βεβαίως κυριαρχεί το θέμα της Ρωσίας και όχι μόνο. Πώς έχει η κατάσταση. Είναι παραμονές της ένταξης της η Ρωσία στον ΠΟΕ. Επίκειται αυτή. Ποια είναι τα εναπομείναντα εμπόδια Στη συνέχεια έχουμε το Μαυροβούνιο. Uh, and Samoa accession... Και άλλες ε, χώρες ε, έχουν ζητήσει να προσχωρήσουν και επίκειται η έγκριση της προσχώρησης από ό,τι έχω καταλάβει. Τρεις περιπτώσεις που γνωρίζω είναι αυτές που σας ανέφερα Τον ε, συνοδεύει και ο κύριος Πολβαρσότη που είναι αναπληρωτής τμήματάρχης και τακτικός επισκέπτης της Επιτροπής μας. Καλώς ορίσατε και πάλι. Κύριε Μπάλας, έχετε το λόγο. Thanks ε, very much, I'm glad to be... Ευχαριστώ. Χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά εδώ για ένα θέμα που ελπίζω ε, σε αυτό το ζωφερό οικονομικό κλίμα το οποίο διατρέχομαι μετά από 18 χρόνια και μιλάω για την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ έχει ε, ε, πιθανότητες να ολοκληρωθεί αυτή. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια σχετικά με τη σημασία ε, αυτής της προσχώρησης της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Η Ρωσία είναι μεγαλύτερη οικονομία που δεν είναι ακόμα μέλος του ΠΟΕ και αυτή η μακρά διαδικασία προσχώρησης είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στις σχέσεις ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία και στην κατάσταση εντός της Ρωσίας επίσης. Ε, λόγω του γεγονότος ότι δεν δεσμεύεται από τις δεσμεύσεις του ΠΟΕ και έχουμε διμερείς σχέσεις με τη Ρωσία που δεν είναι τόσο αποτελεσματικές ε, συμφωνίες ε, ε, σύμπραξης που επηρέασαν αρνητικά την ελευθερία ε, δράσης και είχε επιπτώσεις στις εξαγωγές χρησιμοποιώντας μέτρα SPS, μέτρα υγιεινής. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι το τελευταίο καλοκαίρι χρησιμοποιώντας την δικαιολογία της ε, εστίας ε, μόλυνσης με E. coli σε κάποια μέρη της Γερμανίας είχαν κλείσει εξ ολοκλήρου οι εξαγωγές από όλη για τέσσερις μήνες. Και χωρίς ε, δικαιολογία. Η Ρωσία έχει αυξήσει τους εξαγωγικούς και εισαγωγικούς δασμούς και είναι ελεύθερη να το κάνει. Μέχρι στιγμής ε, έχει, έχει τα... αυτά τα λεγόμενα μέτρα κατά της κρίσης. Ε, δεν υπάρχει όμως κρίση στην ε, Ρωσία όπου παρά τις δυσκολίες κάνει χρήση των ευνοϊκών ενεργειακών τιμών, εξαγωγικών τιμών και είναι σε καλή θέση τουλάχιστον όταν δούμε την οικονομική μεγέθυνση και τις δυνατότητες ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία είναι υπαριθμόν δύο ε, εισαγωγικός εταίρος και υπαριθμόν τρία εξαγωγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε έλλειμμα στο εμπόριο που ε, οφείλεται αποκλειστικά τους στις ψηλές εισαγωγές ε, ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά υπάρχουν προστατευτικά μέτρα της Ρωσίας έτσι ώστε ε, και πάλι σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν σημαντικό και ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, δει την ολοκλήρωση της προσχώρησης της Ρωσίας στην ΠΟΕ. Έχουμε μεταβεί μερικές, ε, μάλλον νομίζαμε ότι θα ολοκληρωνόταν και το 2004 όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε την ε, ε, διαπραγματεύσεις προσχώρησης και υπήρχε ένα πρωτόκολλο για τις διμερείς συμφωνίες. Μετά ακολούθησε μια περίοδος αυξημένου προστατευτισμού από τη Ρωσία και ιδιαίτερα από το 2007 ε, λήφθηκαν μέτρα ε, με νέο δυναμισμό. Το 2007 η Ρωσία ε, θέσπισε μια νέα γεωργική πολιτική που έθεσε τον στόχο να πετύχει 95% αυτάρκεια στα περισσότερα γεωργικά προϊόντα που θέλουν βέβαια να παράγουν περισσότερα. Δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ήθελαν να πετύχουν αυτό τον στόχο, όχι αυξάνοντας την ε, χαμηλή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα της γεωργίας, αλλά αυξάνοντας τον προστατευτισμό τους μέσω των ε, φραγμών των δασμολογικών και μη δασμολογικών. Ε, επίσης, εξαγωγές ξυλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησαν ε, τους, ε, εξαγωγικού δασμού. Ε, είναι ένα πολύ ευνοϊκό εργαλείο της ρωσικής πολιτικής διασφαλίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δίνουν κάποια επιδότηση στην βιομηχανική παραγωγή στη Ρωσία. Οι παραγωγοί παίρνουν τις πρώτε ύλες σε πολύ χαμηλές τιμές και εδώ αναφέρομαι ειδικά στην ενέργεια αλλά σε ό,τι είναι διαθέσιμο σε αυτή την πελώρια χώρα και με τη χρήση των εξαγωγικών ε, επιδοτήσεων μπορούν να αγοράσουν αυτές, ε, αυτές τις πρώτες ύλες σε ψηλότερες τιμές, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη μεταποίηση. Βλέπουμε τον αντίκτυπο αυτής της πολιτικής να επαναλαμβάνεται με επαναλαμβανόμενες ε, στρεβλώσεις της αγοράς έχουμε δει αυτό να επηρεάζει διάφορα προϊόντα όπως ε, το χάλιβα και άλλα γεωργικά προϊόντα. Τελικά, μετά από αυτή τη μακρά διαδικασία, ε, φτάνουμε στην ολοκλήρωση της ε, διαδικασίας προσχώρησης. Και η Ρωσία θα τεθεί υπό κανόνες, διεθνείς κανόνες, και αυτό είναι σημαντικό για μας. Και τα τελευταία 18 χρόνια, ωστόσο, ε, τα αξιοποιήσαμε, διότι αυτό το διάστημα διαπραγματευτήκαμε ε, λεπτομερή δεσμεύσεις με τη Ρωσία. Αυτό το έγγραφο τώρα είναι γύρω στις 800 σελίδες. Είναι σχεδόν έτοιμο και έχουμε μόνο μερικά θέματα τα οποία κρεμούν αυτή τη στιγμή. Ε, με ευτυχής να ανακοινώσω ότι τελικά ε, έχουμε τα τελευταία ε, σημεία στα διμερή θέματα ενώ ε, αυτή τη στιγμή η ρωσική πλευρά δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι η ρωσική κυβέρνηση θα εξετάσει ολόκληρο το πακέτο του ΠΟΕ σύντομα και τότε θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι η συμφωνία για τα διμερή θέματα έχει κλείσει. Τώρα για τις πολυμερείς δεσμεύσεις υπάρχουν ακόμη ορισμένα ανοιχτά ερωτήματα. Το πρώτο είναι η χρήση των ε, μέτρων υγιεινής και φυτοϊγείας είναι εξαιρετική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θέλουμε να έχουμε μια αποτελεσματική πειθαρχία στη χρήση των παρανόμων μέτρων επενδύσεων από άποψη του ΠΟΕ που ε, ε, επιβάλλοντα τοπικού κανόνε ιδιαίτερα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι ένα από τα τελευταία ζητήματα που πρέπει να επιληθούν και εδώ έχουμε ακόμη να ε, αναφέρουμε ότι πρέπει να γίνει κάποια δουλειά στον τομέα των πολυμερών και υπάρχουν κάποια ζητήματα επίσης σχετικά με τις διασφαλίσεις και εγγυήσεις για το πλεόνασμα ε, κρέατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δασμολογικές ποσοστώσεις στο κρέας, ε, τους εξαγωγικούς δασμούς. Θα έλεγα όμως ότι τα περισσότερα θέματα ουσίας τα έχουμε κλείσει. Άρα οι προϋποθέσεις είναι εκεί για, από οικονομικής άποψης για να ολοκληρωθεί η προσχώρηση στον ΠΟΕ. Το σχέδιο το συμφωνηθέν αυτή τη στιγμή είναι να αξιοποιηθεί η ευκαιρία της σύσκεψης της υπουργική του ΠΟΕ στα μέσα του Δεκέμβρη για να καλωσορίσουν την Ρωσία ανάμεσα στα μέλη, το 154ο μέλος του ΠΟΕ, ενώ το Μαυροβούνιο θα έχει την ευκαιρία να προσχωρήσει μάλλον ε, την ίδια χρονική στιγμή. Θα πω και μερικά λόγια γι' αυτό. Είναι κάπως ε, δύσκολο το, το χρονοδιάγραμμα. Δεν έχουμε φτάσει στο τέρμα της διαδικασίας. Έχει ολοκληρωθεί κατά 99%. Παραμένει 1% που όμως παίρνει χρόνο. Πρακτικώς όμως μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες ε, σχετικά με τις ε, δεσμεύσεις για την προσχώρηση της Ρωσίας. Τώρα από οικονομικής άποψης είναι εφικτό. Όμως έχουμε μείζωνα πολιτικά θέματα να επιλύσουμε, να επιλύσουμε το θέμα της ε, διαφοράς ανάμεσα στη Ρωσία και την Γεωργία. Η Γεωργία ως μέλος του ΠΟΕ έχει υποβάλει ε, συγκεκριμένα αιτήματα στη Ρωσία σχετικά με το εμπόριο ανάμεσα στη Ρωσία και τις δύο περιοχές της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Η θέση της Γεωργίας είναι υπάρχουν υποχρεώσεις ε, του ΠΟΕ προς την Ρωσία να παρέχουν παρακολούθηση και επιτήρηση και διεθνείς ε, παρατηρητές ε, εμπορίου σε αυτές τις δύο περιφέρειες που όπως θα γνωρίζετε ε, ε, ανάμεσα ε, στον πόλεμο ανάμεσα στις δύο χώρες αναγνωρίστηκαν ως ανεξάρτητα κράτη. Δεν ακολούθησαν πολλές άλλες αυτό το παράδειγμα, αλλά η Ρωσία θεωρεί αυτές τις δύο περιοχές ως ανεξάρτητες χώρες. με ναι, όλα όσα αυτά, αυτό υπονοεί. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα πολιτικό ζήτημα και ενδυνάμει ε, μια πολιτική αντιπαράθεση. Μελετήσαμε τις απαιτήσει ε, της Γεωργίας και υπάρχει μια αμφιλεγόμενη κατάσταση. Από πολιτικής άποψης η Ευρωπαϊκή Ένωση στεναρά υποστηρίζει την ε, εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και την ανάγκη να επανεγκαθεδρίσει την αυτοκυριαρχία αυτών των δύο περιφερειών που έχουν αποσκιστεί. Όμως ε, δεν βλέπουμε ότι η προσχώρηση στον ΠΟΕ είναι το σωστό φόρουμ για την επίλυση αυτών των βασικών πολιτικών προβλημάτων. Υποστηρίζουμε την τις απαιτήσει της γεωργίας ε, να ε, ακολουθηθεί μια πολιτική διαδικασία αλλά από την άλλη πλευρά δεν ε, θέλουμε να αναμειγνύουμε το εμπόριο με την πολιτική. Οι τρέχουσα θέσεις απέχουν πολύ και παρά αυτό παρά τις προσπάθειες της Ελβετίας να διαμεσολαβήσουν ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτές οι προσπάθειες ε, δεν ήταν πολύ επικοδομητικές μέχρι στιγμής και δυστυχώς υπάρχει πιθανότητα ε, αυτή η ελβετική ε, διαμεσολάβηση να ολοκληρωθεί χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια πολύ δύσκολη επιλογή Δηλαδή πώς να συμφιλιώσουν την πολιτική υποστήριξη προς τη Γεωργία με το μεγάλο μας ενδιαφέρον να δούμε την προσχώρηση της Ρωσίας στην ΕΠΟΕ. Ε, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτή την εξίσωση, αλλά μπορεί να αποφασιστεί τελικά πώς ε, ο στόχος της προσχώρησης της Ρωσίας στον ΠΟΕ φέτος θα μπορούσε να επιτευχθεί. Η ρωσική θέση δεν βοηθάει καθόλου φυσικά. Ακολουθούν μια πολύ σκληροτράχηλη ε, θέση απέναντι στη Γεωργία. Οι σχέσεις ε, τους είναι ανύπαρκτες στην ουσία και δεν έχουν επιδείξει οποιοδήποτε συμβιβασμό από την πλευρά τους. Η Ρωσία επίσης δήλωσε ότι εάν δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία προσχώρησης του ΠΟΕ δεν θα επιδιώξουν περαιτέρω αυτή τη διαδικασία και θα παραμείνουν εκτός του ΠΟΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, θεωρώντας ότι η προσχώρηση ε, στον ΠΟΕ δεν είναι πολύ δημοφιλή στη Ρωσία και ίσως ε, να μην τονίζω και πολύ αυτό το γεγονό. Υπάρχουν δυνατές δυνάμεις στη Ρωσία που δεν θα είναι ικανοποιημένε αν πάρουν τέτοια τροπή τα πράγματα. Ε, αυτό για το οικονομικό μέλλον της Ρωσίας δεν είναι δυνατό να το δουν χωρίς να είναι μέλος του ΠΟΕ και να μην είναι ενσωματωμένοι στην παγκόσμια οικονομία, αλλά είναι ήδη ε, οι Ρώσοι που πρέπει να πάρουν αυτή την απόφαση. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ και σε δύο άλλα θέματα. Ένας από τους παρά, ε, παράγοντες περιπλοκότητας είναι ότι η Ρωσία έχει προβεί σε μια τελωνιακή ένωση με το Καζακστάν. Uh, και με τη Λευκορωσία. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι υπάρχει μια κοινή εμπορική πολιτική με αυτούς τους δύο εμπορικούς εταίρους και αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία δασμολόγησης και για, αυτή, και για αυτές τις δύο χώρες προωθείται. Το Καζακστάν θα προσχωρήσει σχετικά γρήγορα και η Λευκορωσία, η οικονομία της Λευκορωσίας ε, δεν έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές. γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να μην υπάρχει διπλή φορολογία. Εν πάση περιπτώσει, ε, με βάση αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να προσχωρήσουν στον ΠΟΕ. Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο θέμα που θα μπορούσε να μας απασχολήσει και ως προς το Μαυροβούνιο η προσχώρηση αυτή θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια. Υπάρχει μία χώρα, η Ουκρανία, η οποία δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με αυτή τη μικρή χώρα, γι' αυτό και δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ελπίζουμε όμως και σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα να επέλθει ένα συμβασμός ανάμεσα στις δύο χώρες και το Μαυροβούνιο να γίνει μέλος του ΠΟΕ. Το γεγονός ότι η Ουκρανία όμως μπορεί να παρατείνει αυτή την αβεβαιότητα ως προς την προσχώρηση δείχνει ότι δεν πρέπει να υποβιβάζουμε και το θέμα της γεωργίας γιατί η Γεωργία έχει προβάλει βέτο. Θα σταματήσω εδώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Ο συνάδελφός μου, ο Πάολο, μπορεί να σας ε, να σχολιάσει περαιτέρω. Και βεβαίως θα ακούσω και τα σχόλια των μελών της Ίντα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εκτενή παρουσίωση Ας αρχίσουμε με τον Ρόμπερτ Στέρτ, ο οποίος είναι εδώ και είναι και ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ, Πίτερ, για αυτή την εισβάθο συζήτηση. Και αυτό που με απασχόλησε είναι μερικά από τα σημεία που έθιξες όταν είπες ότι είμαστε κοντά σε μια διμερή συμφωνία. Είπες αρχικά ότι θα την έχουμε φέτος. Όμως στη συνέχεια είπες ότι ίσως υπάρχουν προβλήματα με τη Λευκορωσία και άλλες χώρες που θα αναχαιτήσουν τη διαδικασία. Μπορεί να το κάνει αυτό και η Γεωργία. Μπορείς να μας πεις τι εννοείς ότι είμαστε κοντά στη διμερή συμφωνία. είπε επίσης ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε την πολιτική με το εμπόριο, μα είναι αλληλένδετες αυτές οι σχέσεις, σωστά ή λανθασμένε. Όσο καιρό βρίσκομαι εδώ αυτό διαπιστώνω. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοούσες. θα παρακολουθήσω την απάντηση. Αυτά είναι θέματα ελάσσονα ζητήματα. Σκιώδης. Σόλτς από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω. Ήταν πάρα πολύ πλήρης, εξαντλητική η παρουσίασή σας της ε, σημερινής κατάστασης των ε, πραγμάτων στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ, κυρίως για τη Ρωσία. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την τελωνιακή τους ένωση με τη Λευκορωσία και το Καζαχστάν. Τι σημαίνει αυτό, εάν προσχωρήσει η Ρωσία. Αν ολοκληρώσει επιτυχώς, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι τα τέλη του έτους της διαπραγματεύσεις και μπει. Τι θα σημαίνει αυτό για τα προϊόντα από τις χώρες αυτές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έτσι, εισαγωγές, εξαγωγές και τα λοιπά από το Καζαχστάν και τη Λευκορωσία. Και τι σημαίνει αυτό επίσης προς το παρόν. Θα, θα ανοίξει προοπτική να ε, προσχωρήσουν στον ΠΟΕ και το Καζαχστάν και η Λευκορωσία ή θα είναι ένας τρόπος να δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε να τους φέρουμε και εκείνους στον ΠΟΕ και να δώσουμε στη Ρωσία να καταλάβει τι μπορεί να, να ε, συνεισφέρει ως μέλος του ΠΟΕ. Επιπλέον, έχετε τίποτα ενδείξεις ή και αποδείξεις από τη ρωσική πλευρά ή και από άλλες πλευρές για το γύρο της Δόχα στον ΠΟΕ και ποια είναι η θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την ολοκλήρωση του γύρου της Δόχα. Ο Γιάννικ Ζαντο από τους Πρασίνους. Ε, ένα σχόλιο μόνο. Εμιδίασα λίγο όταν είπατε να μην αναμειγνύουμε την πολιτική με το εμπόριο. Ενδιαφέρον μου φαίνεται αυτό, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τη Ρωσία, όπου κανείς ασκεί πολιτική ελέγχοντας την οικονομία. Πλουτίζει, κυβερνάει και ελέγχει την οικονομία. Γιατί αν υπάρχει μια χώρα που η πολιτική και η οικονομία είναι τόσο διαπεπλεγμένες, η χώρα αυτή είναι η Ρωσία. Και επιπλέον, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε ο Ρόμπερτ, ε, θα πρέπει να ε, το δεχτούμε αυτό ότι και στις εμπορικές συμφωνίες στη διαπραγμάτευση πολιτική είναι. Σε αυτό το πνεύμα είμαστε. Ας μην προσποιούμαστε ότι δεν κάνουμε πολιτική. Αλλιώς δεν προχωρούμε με αυτά τα μισόλογα. Σαν να πηγαίνετε στην Ελλάδα τώρα να δώσετε μια διάλεξη στην Αθήνα και να λέτε στους Έλληνες πολίτες ότι η οικονομία και η πολιτική α, είναι δύο πράγματα τελείως ε, χωριστά και να μην τα αναμεγνύεται. Μα το εμπόριο και η οικονομία πάνω απ' όλα είναι πολιτική και στη σχέση μας με τη Ρωσία είναι και ένα σύστημα τόσο διεφθαρμένο και διεστραμμένο που πραγματικά πρέπει να κάνεις και πολιτική εκεί. Ευχαριστώ. Δεν ζητεί κανείς άλλο το λόγο. Έχετε πάλι εσείς για να απαντήσετε στα σχόλια, στα ε, θέματα που σας έθεσαν υπόψη, στις ερωτήσεις, αν θέλετε και ο κύριος Καρσότη. Ναι, βλέπω ότι αυτά που είπα, που θα έπρεπε να είχα πει, ότι η πολιτική και η προσχώρηση στον ΠΟΕ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι, διότι ο ΠΟΕ είναι μια διεθνής οργάνωση, ένας οργανισμός που ρυθμίζει το εμπόριο. Εγώ σέβομαι την άποψή σας. Αλλά πιστεύετε ότι μπορεί να επιληθεί ένα θέμα εδαφικής ε, διένεξης Γεωργίας-Ρωσίας στα πλαίσια του ΠΟΕ, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτό. Και μάλιστα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για την προσχώρηση στον ΠΟΕ. Πρόκειται για στρατιωτική κατοχή αυτών των ε, επικρατιών ε, από τη Ρωσία ε, που είναι κάτι για το οποίο εκφράζουμε τη λύπη μας και μάλιστα πάρα πολύ έντονα. Ελέγχουν κάθε ζωή στη περιφέρεια και κρατούν στην εξουσία καθεστώτα τα οποία μπορεί κανείς να έχει διαφορετική αντίληψη για το κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται. Αλλά αυτά τα ε, ζητήματα δεν λύνονται εν ώψη της προσχώρησης μιας χώρας στον ΠΟΕ, όπου έχει να κάνει με ε, ειδικά ζητήματα και ανησυχίες εμπορίου. Δεν υπάρχει πουθενά λέξη στον ΠΟΕ που να ε, βάζει πολιτικούς όρους για να γίνεις μέλος. Εσείς μπορεί να διαφωνείτε ότι δεν είναι σωστή η προσέγγιση, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση και τα συστήματα σε χώρες που είναι μέλη του ΠΟΕ. Και επίσης ο ΠΟΕ κοιτά την οικονομική πολιτική και την εμπορική πολιτική και κατά πόσο αυτή είναι συμβατή με τους πολυμερείς κανόνες που έχουν αποφασίσει τα μέλη. Και τα μέλη τότε αποφασίζουν αν θα ενταχθεί ή όχι. Βεβαίως έχει δικαίωμα κάθε μέλος του ΠΟΕ uh, ε, γιατί λειτουργεί συνενετικά Λοιπόν, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να βάζει πολιτικά προαπαιτούμενα για να δώσει το ok ε, στην προσχώρηση μιας νέας χώρας. Ε, αυτό εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλούμαστε να το κρίνουμε, εάν εξυπηρετεί ή όχι τα συμφέροντα της Ένωσης. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι ε, από πλευράς οικονομικής και συστημικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση το να είναι η Ρωσία εντός του ΠΟΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα ποια θα είναι η πολιτική απόφαση του Κοινοβουλίου σας των κρατών μελών. Ότι θα πρέπει να λυθεί η εδαφική διαφορά που έχουν οι δύο χώρες. Ε, τότε η Ρωσία δεν πρόκειται να μπει στο προσεχές μέλλον. Είναι γεγονός αυτό, δεδομένη την κατάσταση. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, αυτή είναι η δυνατότητα. Εγώ εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου εδώ. Νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί τα ευρύτερα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι δική μου υπόθεση αυτό το να κρίνω. Εσείς καλείστε να το κρίνετε και ε, μπορεί η πρόταση ε, αυτή, η πίεση αυτή να βρεθεί πολύ γρήγορα μπροστά σας. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα περιβαλλοντικά, πρότυπα εργασιακά που είναι κοντά σε θέματα εμπορίου, βεβαίως. Αλλά ο έλεγχος ε, ενός εδάφους με κάθε σεβασμό δεν συνδέεται πάρα πολύ με το εμπόριο ούτε άμεσα. Μπορεί να είναι πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα, μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικό ειδικά για τη γεωργία και το σεβόμαστε, αλλά αν αυτή η εδαφική διένεξη λυθεί ή όχι δεν μπορεί να είναι ε, προαπαιτούμενο ούτε να επηρεάζει τις συνθήκες ε, δημιουργίας οικονομικής συνεργασίας με τη Ρωσία. Για να πω και κάτι ακόμα, έχετε απολύτως δίκιο όταν αναφέρεστε στην οικονομική κατάσταση και την οικονομική πολιτική της Ρωσίας. Ότι είναι πολιτικές αποφάσεις και εμπορικές. Αλλά μπαίνοντας στον ΠΟΕ, αυτό περιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν λέω ότι τερματίζεται. Περιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, Αναλαμβάνοντα διεθνεί δεσμεύσει, η Ρωσία δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει τι σημερινέ πρακτικέ. Ε, ε, αυξάνει ε, τους δασμούς και τα μέτρα SPS, διότι θα έχει δεσμευτεί διεθνώς και θα πρέπει να τηρεί αυτές τις συμφωνίες θα είναι εύκολο ε, ο μέλος του ΠΟΕ. Όχι, σίγουρα, όχι, ούτε εκείνα είναι. Και είπε κανείς ότι ήταν σφάλμα η προσχώρηση της Κίνας στον ΠΟΕ. Όχι, δεν νομίζω. Γι' αυτό ισχύει και για τη Ρωσία. Τους φίλους τους διαλέγεις, του γείτονέ σου, όχι. Αυτή είναι η Ρωσία, είναι γείτονά μας και είμαστε υποχρεωμένοι να τη δεχθούμε όπως είναι. και να συμβιβαστούμε με αυτή την πραγματικότητα, να συνεργαστούμε με αυτή τη χώρα και να σε εκτιμήσουμε τουλάχιστον ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πολιτική βούληση παρά την ισχυρή αντίσταση πολλών κλάδων και εντός της Ρωσίας. Η ηγεσία της χώρας φαίνεται ότι έχει καταλάβει και αναγνωρίσει ότι είναι και προς το δικό τους μακροπρόθεσμο συμφέρον να ενταχθούν στον ΠΟΕ. Για να έρθω τώρα για Ε, τις διμερείς ε, ε, συνομιλίες υπό όρους έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις αλλά περιμένουμε την επιβεβαίωση της ρωσικής κυβέρνησης Πάντως είμαι βέβαιος σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι Ορισμένα ζητήματα που εκκρεμούν και λεπτομέρειες μπορούν να λυθούν ε, τις ερχόμενες εβδομάδες. Η αβεβαιότητα και ο αστάθμητος παράγων τελικά είναι η γεωργία. Ε, Για να αποφασίσει και θα καθορίσει αν θα μπει η Ρωσία στον ΠΟΗ ή όχι. Η Τελωνιακή Ένωση έχει κάποιο χαρακτήρα έτσι που διαταράσει ε, την προσχώρησή Έτσι. Αν δεν είχε τελωνιακή ένωση, ενδεχομένως η Ρωσία να ήταν ήδη μέλος στον ΠΟΕ. Τι σημαίνει αυτή η τελωνιακή ένωση. Καλείται η Ρωσία να ευθυγραμμίσει ε, την πολιτική της στα πλαίσια του ΠΟΕ και απέναντι στους δύο εταίρους της Τελωνιακής της Ένωσης. Ζητήσαμε και λάβαμε πάντως νομική εξασφάλιση ε, και εγγύηση από τη Ρωσία ότι ό,τι ε, αναλάβει ως δέσμευση ε, στον ΠΟΕ θα εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες δύο χώρες. Έχει συναυθεί αυτή η συμφωνία και μεταξύ των τριών μερών της Τελωνιακής Ένωσης. Είναι σε διαδικασία κύρωσης. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε θα επιμείνουν να ισχύσει αυτό. ήταν πάρα πολύ εύκολο να παίζουν διάφορα παιχνίδια εκεί και να. Ε, έχουμε προβλήματα με τις δύο χώρες αυτές της Θελωνιακής Ένωσης. Τι σημαίνει η προσχώρηση. Ο κοινός δασμός θα πέσει σε επίπεδο ε, που θα έχουμε διαπραγματευτεί με τη Ρωσία, δηλαδή εξαγωγές της ευρωπαϊκή Ένωσης και προς τη Ρωσία και προς τη Λευκορωσία και στο Καζαχστάν θα διευκολύνονται ε, και τα, άλλα μέτρα, τα μη δασμολογικά, ε, θέματα υγείας, τεχνικά θα ισχύουν και στην επικράτεια της Τελωνιακή Ένωσης. And Ελεύθερη κυκλοφορία λοιπόν και στις τρεις χώρες, όπως και στην εσωτερική αγορά ισχύει και ε, οπωσδήποτε η Τελωνιακή Ένωση βασίζεται στο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πολύ μεγάλη ήδη ολοκλήρωση. Αν προσχωρήσουν στον ΠΟΕ θα χρειαστεί διαπραγμάτευση με τη σειρά τους. Το Καζαχστάν ήδη έχει ορίσει, μάλιστα έχει υπογράψει ε, τελωνιακές ε, συμφωνίες και έχει έρθει και ο αρμόδιος ε, Καζάκος υπουργό αυτό τον καιρό εδώ και διαπραγματευόμαστε για τις εξαγωγικές επιδοτήσεις. Αυτό έχει να κάνει με τις πρώτες ύλε και την ενέργεια και την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πάρα πολύ σημαντικό. Και μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις με το Καζαχστάν, μπορεί γρήγορα να ενταχθεί. Δύο λεπτά έχετε ακόμα, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις και θα σταματήσω εδώ. Χελμούτ Σόλτς, θέλεις να ξαμιλήσεις. Ναι. Μια πολύ σύντομη συμπληρωματική ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, αλλά πολύ σύντομη αναμένεται οι εκλογές του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου στη Ρωσική Ομοσπονδία να μας δώσουν μια καλύτερη διαπραγματευτική θέση για να καταλήξουμε με τη Ρωσία ή θα υπάρχουν τίποτα προβλήματα εκεί. Of course, uh, of course, never... Θα αλλάξει κάτι. Δεν μπορούν να γίνουν τέτοιες προβλέψεις, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω ότι θα διευκολύνονταν τα πράγματα με πρόεδρο Πούτιν, πρωθυπουργό Πούτιν. Έχουν συμφωνηθεί οι όροι με τη Ρωσία η όροι προσχώρησης κατά 99% κανένας δεν θέλει να ξανανοίξει αυτό το κεφάλαιο νομίζουμε ότι θα είναι ιδιαίτερα πλεονεκτική για τους ετερους τους οικονομικούς εταίρους της Ρωσίας και το θέμα που έχει σημασία είναι να επιληθεί η διένεξη Γεωργίας και Ρωσίας. Ευχαριστούμε τον Πίτερ Πάλας που εμπλούτησε τις γνώσεις μας σε θέματα προσχώρησης της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Θα ξανασυνεδριάσουμε στις 22-23 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.